Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης με δύο τροποποιήσεις, αν συμφωνείτε. Μετά από το σημείο 7, μία επιστολή Euh, να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε σε αίθουσα συνεδρία της Επιτροπής και να αποφεύγονται οι προσωπικές συζητήσεις, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, μετά το σημείο 7 αν συμφωνείτε θα εγκρίνουμε μια επιστολή για την κινητοποίηση του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αιτήματο τη Ιταλία για την περιοχή Τρεντίνο Άλτο. Είναι επίγουσα περίπτωση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μπορούμε να το δεχθούμε. Και στο σημείο 13 για την ψηφοφορία για την γνωμοδότηση για κονσάρι για τι συνθήκε ε, εισόδου και παραμονή υπηκόνων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ε, ενδοεπιχειρησιακών αποσπάσεων. Αυτή η ψηφοφορία μεταφέρεται στην επόμενη συνεδρίαση και αντί αυτού του σημείου θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Σέργιο Κοφεράτη όπως έχει ήδη προβλεφθεί. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρούμε ότι τροποποιήθηκε η μέση διάταξη και εγκρίνεται. Στο σημείο 2 η Πρόεδρος έχει κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχήν θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας ε, αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο. Έχουμε web streaming. Πρέπει να σας πληροφορήσω κάτι το οποίο εσείς ήδη το γνωρίζετε, ότι για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ, ένα θέμα που είναι ε, θεμελιώδες για μας, η οδηγία δηλαδή για τον χρόνο εργασίας, η κοινωνική εταίρη άνοιξαν τις διαπραγματεύσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν εννέα μήνες για να καταλήξουν σε συμφωνία. Πριν δούμε περί τίνος πρόκειται, όπως συμφωνήσαμε στη συνεδρία της συντονιστών, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις διαπραγματεύσεις τους και πώς να έχουμε επαφή με τους μεν και τους δε. Τελευταία παρατήρηση, θέλω να σας συστήσω τον κύριο Ρομπέρ Σεπόλτ, που είναι καινούριο στην γραμματεία της Επιτροπής Απασχόλησης. Ήταν υπάλληλο της Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Είναι νομικός, ειδικό στα θέματα συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. θα έχει επομένως ε, άπλετο χώρο να αναπτύξει τα ενδιαφέροντά του στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε. Vous allez utilement... Θα ενισχύσετε ε, το, την ανδρική ποσόστοση των μελών της γραμματείας μας. Λοιπόν, στο σημείο 3 Στο σημείο 3 της μείσια διάταξης έχουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007-2012 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες που θα μας παρουσιάσει η συγκήτρια, η κυρία Καϊμά Ντελή. Αλλά πριν της δώσουμε το λόγο, θέλω να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής μας και ιδιαίτερα τους συντονιστές ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. βλέπω τα στρατηγικά ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς στην Επιτροπή μας μέσα στους προσεχείς μήνες και σαφώς αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι μία από τις προτεραιότητες δεδομένης της γενικής λιτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δίνω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Voilà, pardon. Euh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 27 συμβιβαστικές τροπολογίες που πραγματικά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μου. Είμαι ικανοποιημένη από το σύνολο των συμβιβασμών. Ε, ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν με ενθουσιασμό για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που θα μας επιτρέπει από αύριο να νιώθουμε περήφανοι για την έκθεση αυτή. Μιλάμε βέβαια για ένα πρώτο βήμα, δεδομένου ότι πρόκειται για μια ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα δούμε αν θα υπάρξει άλλη ευρωπαϊκή στρατηγική τα επόμενα έτη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να τους ευχαριστήσω θερμότατα και τους ίδιους και τους βοηθούς τους γιατί υλοποίησαν αυτά τα οποία από χρόνια ζητούν οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι τον ε, διάλογο, ε, κοινωνικό διάλογο για τα θέματα των επαγγελματικών ε, ασθενειών και για να φροντίσουμε ώστε στο μέλλον κανένας να μην πάσχει από ασθένειες ή ατυχήματα που να οφείλονται στην εργασία του. Ελπίζω ότι το σύνολο της, ε, των της Επιτροπής θα ψηφίσει τους συμβιβασμούς αυτούς και όλες τις τροπολογίες και θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέρφων σε δύο συγκεκριμένες τροπολογίες. Η 148 η οποία έχει σκοπό τη δημιουργία μιας πραγματικά ανώτατης ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σεβασμού της Εργασίας που θα ασχοληθεί με τα θέματα των αποσπασμένων εργαζομένων και οι οποίοι πρέπει να καλύπτονται από την νομοθεσία, όπως επίσης και την τροπολογία που ε, αφορά αυτούς που εργάζονται σε υπεργολαβία. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ο σκιώδης εισηγητής, ο κ. Κράιτσμαν, ε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί είχε οργανώσει μια ακρόαση και μου ζήτησε να θέσω κάποια θέματα. Η συζήτηση για την έκθεση αυτή ήταν εντατική τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως επειδή ασχολείται με τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα. Πρέπει να γίνουν πράγματα σε διάφορους τομείς. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεί ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και ότι μερικά προβλήματα είναι καλύτερα να λυθούν σε εθνικό επίπεδο. Οι διάφορες ε, οι διάφοροι συμβιβασμοί επιλύουν τις ανησυχίες της Επιτροπής και χαιρόμαστε που έχουμε φτάσει σε λογικές λύσεις στα περισσότερα ζητήματα. Παραδείγματο χάρη λαμβάνονται υπόψη οι δικές μας απόψεις σε άλλους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για να μπορέσουν να τεθούν σωστές προτεραιότητες στο μέλλον. Τώρα, εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα με τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών. Γιατί ενώ υπάρχουν ενδεχόμενοι κίνδυνοι, του οποίου αναγνωρίζουμε, δεν ε, εμπλεκόμαστε σε συγκεκριμένε περιπτώσεις, στην προκειμένη περίπτωση είναι ανατεχνολογία. Επίσης, όσον αφορά την πρόληψη, θα προτιμούσαμε να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα μέτρα που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους. Χαίρομαι για τον συμβιβασμό ε, τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ε, για την κάλυψη των εργαζομένων από επαγγελματικέ ασθένειε και χαίρομαι επίση που υπάρχει ε, συγκεκριμένο θέμα για τον ε, blacklist αυτών των εργαζομένων. Ε, αυτό που χρειάζεται σε πολλούς τομείς δεν είναι νέα νομοθεσία αλλά η καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθεσιών και θελουσίες ε, συμφωνίες. Επίσης μου ζήτησαν να, ευχαριστήσω ιδιαίτερως την εισηγήτρια αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους σχεώδεις για τις παραγωγικές συζητήσεις των τελευταίων εβδομάδων και την θέλησή τους να καταλήξουν σε συμβιβασμού σε τόσα πολλά θέματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω καλά νέα και κακά νέα. Ε, τα καλά νέα θα πω πρώτα και μετά τα άσχημα. Τα καλά νέα είναι ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Είχαμε ένα εξαιρετικό κείμενο βάσης από την Κάρη Μαντελή και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία βουλευτές, βοηθοί και γραμματείες και αυτό είναι ελπιδοφόρο για τον τρόπο που εργάζεται το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι ελπιδοφόρο για την ευρώπη και τους πολίτες της. καταφέραμε και φτάσαμε σε εξαιρετικούς συμβιβασμούς έχοντας στο μυαλό μας την υγεία και την ασφάλεια των ευρωπαίων εργαζομένων. αυτά είναι τα καλά νέα. τα κακά νέα είναι ότι αυτό το θεωρητικό κείμενο το οποίο υιοθετούμε εμείς εδώ θα πρέπει η Κομισιόν να πάρει την πρωτοβουλία να το περπατήσει, να το κάνει πράξη, να το βάλει μέσα στη ζωή. Και τα νέα, οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι η Επιτροπή αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που αποφασίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων δεν σκέπτεται να τα ε, να τα επενδύσει με μία νομοθετικού τύπου κίνηση. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η έκθεση γίνεται ακόμα πιο σημαντική, γι' αυτό ακριβώς ο τρόπος που εργαστήκαμε αποκτάει ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να πιέσουμε σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να πιέσουμε την Επιτροπή να λάβει υπόψη της σοβαρά και να ενεργήσει στην πράξη τα δέοντα για το θέμα της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών στην εργασία τους. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για παρόμοια θέματα να έχουμε μόνο καλά νέα. Σας ευχαριστώ. Δεν, δεν βλέπω κανένας άλλος να ζητάει το λόγο. Α, ο κύριος Μπέκερ. Δεν μπορούσε να παρόν ο κύριος Μπαχ για λόγους υγείας και ζητά συγγνώμη. Μου ζήτησε εκ μέρους του να σας διαβάσω την εξή θέση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελή για την καλή συνεργασία με την καλή συνεργασία των σχεδόν εισηγητών καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε 26 τροπολογίες οι οποίες ικανοποιούν όλους. Το θέμα της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας μας αφορά όλους και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων και να την προσαρμόζουμε στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις μας και για ιατρικά ζητήματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτή η έκθεση θα συνεισφέρει στην επόμενη στρατηγική, η οποία θα είναι εξίσου, ε, εξίσου ικανοποιητική όσο και η προηγούμενη και έχω και μία προσθήκη που δεν συμπεριλαμβάνεται στο γραπτό κείμενο που σας διάβασα από τον κύριο Μπαχ και συγκεκριμένα ε, στα θέματα ε, της υπεργολαβίας ε, δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Αυτό συμπλήρωση το αναφέρω. Uh, uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Καρίμα Αντελή για τις, ε, γιατί και τις προτάσεις μου για συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες πιστεύω όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να καταλήξουμε σε, ε, στις συμβαστικές αυτές τροπολογίες για τα επιστημονικά δεδομένα οι επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα πρέπει να μιλάμε για ενημερωμένα δεδομένα Τώρα, Υπάρχουν ήδη οδηγίες για τα μαγνητικά πεδία που θα συζητηθούν και αύριο. Ε, για να σας πω ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα της Κομισιόν κάποιες προτάσεις και καταλαβαίνω βέβαια και τις δικές σας παρατηρήσεις. Ούτως ή άλλως πρόκειται για οδηγίες που ήδη ε, συζητώνται και είναι οδηγίες ε, κλειδιά. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν ζητά... Α, ο κύριος Σαρκάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Ράπτη η σοσιαλίστρια βουλευτής μίλησε για μία φήμη η οποία κυκλοφορεί που λέει ότι η Κομισιό αυτούς τους καιρούς ε, κρίσης ε, που περνάμε ε, δεν σκέφτεται να λάβει μέτρα για την στρατηγική στο χώρο εργασίας. Εάν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε η έκθεση της κυρίας Ντελή και ό,τι άλλο έχουμε κάνει θα ήταν μια αποτυχία. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, υπάλληλοι της Κομισιόν εδώ στην αίθουσα και θα ήθελα να μας πούνε ξεκάθαρα τι πρόκειται να γίνει. Θα πρέπει να πούμε τις απόψεις μας σαν κοινοβούλιο και θα πρέπει και η Κομισιόν να γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η σοσιαλιστική ομάδα δεν θα ήθελε όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε να μείνει στα χαρτιά και να είναι μια άσκηση γραφειοκρατίας. Από πλευρά της Κομισιόν, μήπω κάποιο από του παρατηρητέ ίσω ε, κάποιο από την πλευρά τη Κομισιόν θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριε Κλάρκ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος, κύριε, Κλάρκ, θέλετε να πάρετε μέρος στη συζήτηση. Α, έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δύο ερωτήσεις για δύο διαφορετικές τροπολογίες. Η πρώτη, η τροπολογία 213 του Τόμας Μάνα, που ζητάει για την ότι θα πρέπει να περιοριστεί και η εργασία την Κυριακή, όπως και η νυχτερινή εργασία, ας πούμε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Κομισιόν στο γεγονός ότι αυτά ακούγονται καλά μεν, η ανάπαυση την Κυριακή κτλ. Παρόλα αυτά πάρα πολλές ε, δουλειές ε, κάνουν πολύ, ε, πολλές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις κάνουν πολλή δουλειά την Κυριακή και αν τους απαγορευτεί να ανοίγουν την Κυριακή θα έχουν μεγάλη ζημιά και κυρίως τώρα που με την κρίση που περνάμε χρειάζονται και το τελευταίο ευρώ και το τελευταίο πένι. Επίση ή άλλο τροπολογία 171. Όπου θέλει να διαγράψει την τροπολογία που λέει, ζητάμε από την επιτροπή να προτείνει μια οδηγία, η άλλη τροπολογία 171 όπου θέλει να διαγράψει την τροπολογία που λέει ζητάμε από την Επιτραπή να, προβά, να προτείνει μια οδηγία η οποία ε, μια πρόταση οδηγία που θα προστατεύει την εγρήγορηση και την επιγνωμοσύνη τη περιπτώσει ατόμων που ανησυχούν εύλογα για του κινδύνου οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν στο πλαίσιο μια επιχείρηση. Κοιτάξτε, εδώ καρφώνουμε. Και risks and the like to their employers or to... Τι θέλουμε να κάνουμε. Ε, θέλουμε να, τους, ε, να σταματήσουμε να πνίξουμε. Δεν, δεν πρέπει να πνίξουμε αυτούς ε, που προσπαθούν να μας ενημερώσουν και να, να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο γιατί ο κύριο Μπέκερς ε, μίλησε εκ μέρους του ΕΛΚ και εκ μέρους του Ζορς Μπαχ. Προσωπικά ε, θα ήθελα να πω στην Καρίμα Δελή πόσο πολύ εκτιμήσαμε το γεγονός ότι μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε μαζί τις τροπολογίες αυτό το ανοιχτό πνεύμα που έδειξε και το πνεύμα ε, συνεργασίας που επεσήμανε και η κυρία Ράπτη είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το ζήτημα. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή ε, προετοιμάζονται συμπληρωματικές οδηγίες οι οποίες δεν θα μπορέσουν όλες να μπουν στο κείμενο αυτό και στην έκθεση για την υγεία των εργαζομένων και συγκεκριμένα την υγεία των εργαζομένων που υπόκεινται στην ηλεκτρομαγνητική, ε, στα ηλεκτρομαγνητικά κείμενα ε, κύματα, με συγχωρείτε, ε, θα είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της έκθεσης. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτό το πεδίο, αν μου επιτρέπετε, στις πολύ συγκεκριμένες οδηγίες και να προσπαθήσουμε να μην εμποδίσουμε τις οποιαδήποτε απαραίτητες εξελίξεις. Ήδη, κυρία Πρόεδρε, ξεπερνάμε μόλις ε, μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την ε, οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ναι, καταλαβαίνω συνάδελφε την ανησυχία σας για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να ακούσουμε τις ε, εξηγήσει της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Ανεξάρτητα από τα από τα θέματα των διαφόρων κειμένων, ε, η Κομισιόν, και εδώ συμφωνούμε όλοι μας, ε, θα πρέπει να μας πει τι προτίθεται να κάνει ε, με κάποια ζητήματα τα οποία είναι, αποτελούν με μεγάλη προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής και που δεν θα ήθελα να εγκαταλείψουμε. Λοιπόν, θέλετε να πάρετε το λόγο εξ ονόματος της Κομισιόν για να απαντήσετε σε αυτές τις ανησυχίες μας και αν έχετε να προσθέσετε για κάτι ε, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, όχι να μας πείτε την άποψή σας, αλλά να συμπληρώσετε κάποια κενά, αν θέλετε, που μπορεί να υπάρχουν και να μας πείτε και κάποιες ε, ενδείξεις για αυτό το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ε, φήμη ε, σχετικά με τις προθέσεις του Προέδρου της Επιτροπής ε, για το, για το τι θα γίνει με τα κείμενα αυτά. Από ό,τι ξέρω, το πρόγραμμα των εργασίας του 2012 έχει οδετηθεί και εκεί προ προβλέπετε να προετοιμάσουμε την στρατηγική η οποία θα ακολουθήσει αυτή την οποία αναθεωρούμε τώρα, δηλαδή και ε, η, έκθεση, η ενδιάμεση έκθεση θα χρησιμοποιηθεί όπως και άλλα στοιχεία για να ε, τροφοδοτήσουμε την, ε, τις εργασίες μας για τη νέα στρατηγική. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω αυτές τις φήμες, μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε όπου προέρχονται, αλλά το μόνο το οποίο θα ήθελα να σας πω αυτή τη στιγμή η εξ ονόματος της Κομισιό είναι ποιο είναι το πρόγραμμα εργασία το οποίο προτίθεται να υιοθετήσει η Κομισιό μετά από, την, ε, από τις συζητήσεις που είχαμε και με το Κοινοβούλιο. Η κυρία Ντελή έχει το λόγο. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο βασικά θέματα. Καταρχάς μιλήσαμε για την υπεργολαβία και να σας πω ότι το πρόβλημα αυτό είναι σημαντικό και αναφέρεται και στην τροπολογία 48 που θα ήθελα να υπερψηφιστεί αύριο. Επίσης, ο κύριος Μπέκερ είπε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε όλα τα άτομα τα οποία στις επιχειρήσεις τους αντιμετωπίζουν τους ε, ανωτέρους τους που θέλουν να τους ε, ε, ε, να θέλουν να προστατεύσουν την υγεία τους κτλ. Ούτως ή άλλως η τροπολογία αυτή έχει σαν στόχο αυτό ακριβώς τα πράγματα και θα ήθελα να, το, να σας το υπενθυμίσω αυτό και να το διευκρινίσουμε. Είναι η συμβιβαστική πρόταση ΤΕ που είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε και εσείς πρέπει να προστατεύσουν αυτά τα άτομα τα οποία φροντίζουν αν θέλετε και κρούν τον κόμιο του κινδύνου. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ε, κύριοι συνάδελφοι ότι εδώ σε αυτή την ε, ενδιάμεση έκθεση δεν πρόκειται να εγκαταλείψω αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει Θέλω να καταλήξουμε σε μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για τις συνθήκες εργασίας, γιατί δεν είναι απλώς μια ανάγκη αυτό, είναι ε, κατεπήγον το θέμα. Και θα είμαι πραγματικά, θα επαγρυπνώ και θα βλέπω ακριβώς τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε με το σημείο αυτό. Θα ψηφίσουμε αύριο. Τώρα, περνάμε στο σημείο 4, ε, στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, εισηγητής ο κύριος Σβέν Γκίγκολντ. Τι έχετε να μας πείτε όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων. Να μας πείτε, να μας παρουσιάσετε τα συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ πρόκειται για συζήτηση των τροπολογιών. Δεν χρειάζεται να σας τις παρουσιάσω λοιπόν λεπτομερώς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, διότι κάναμε μια πολύ καλή συνεδρίαση. Υπάρχει και το νέο μέλος της ομάδας των Πρασίνων που δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να μπει με τους ε, πράσινους ή με το ίσια με τον κύριο Σόγκο και με την Νάντια Χίρς και τον κύριο Χέρμαν, με όλους τους κοιοδησίτες. Είχαμε πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Και τουλάχιστον έχουμε τώρα συμβαστικέ τροπολογίε, τι οποίε να μπορούν τουλάχιστον οι τέσσερι ομάδε να συμφωνήσουν. Και Χέρμαν, φαντάζομαι ότι είχατε κάποια προβλήματα με κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε. Υπάρχει ευρεία συμφωνία για να υποστηρίξουμε την κοινωνική αλληλεγγύη στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων στον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό, αλλά και γενικότερα. Ίσως να θυμάσαι ότι την περασμένη εβδομάδα έγινε μια ευρεία διάσκεψη που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του κυρίου Μπαρόζο, του κυρίου Νταλή και του κυρίου Μπαχνιέ, με πάνω από 800 συμμετέχοντες από τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της ε, ε, οικονομίας της αλληλεγγύης. Πολύ καλό μήνυμα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα νέο πνεύμα προθυμίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουν περισσότερο και η έκθεσή μας με τις συστάσεις τις οποίες κάνουμε φτάνει την κατάλληλη στιγμή. Υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την κοινωνική οικονομία που ήδη συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην σταθερότερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμβαστικές λύσεις λοιπόν πιστεύω ότι είναι καλές. Δεν είχαμε πρόβλημα να καταλήξουμε σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Κρατήσαμε τη βασική εικόνα της έκθεσης. Είναι πιο ισορροπημένη τώρα η έκθεση με αυτές τις τροπολογίες. και περισσότερο θα ήθελα να ακούσω τα δικά σας σχόλια τώρα παρά να σας παρουσιάσω αυτές τις τροπολογίες που λίγο πολύ τις ξέρετε και ίσως και οι σκιώδεις συζητητές θέλουν να λάβουν το λόγο. Πραγματικά πιστεύω ότι η έκθεση αυτή φτάνει την κατάλληλη στιγμή και προσβλέπω και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής αν μπορούμε να δώσουμε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε τη γνώμη της Επιτροπής για τις συστάσεις που θα προκύψουν από την έκθεση. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη της Επιτροπής. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Νάντια Χιούς δεν είναι σήμερα που είναι σκιώδης εισηγήτρια και μου ζήτησε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την αφοσίωσή του και για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό και για την πολύ καλή δουλειά που έκανε για τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Τις υποστηρίζει όλες και πιστεύει ότι στέλνουν θετικά μηνύματα προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κυρία Χέγνε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι συνεργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά και νομίζω ότι όλοι κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό και οι συμβαστικές τροπολογίες είναι επικοδομητικές και μας είναι αποδεκτές. Πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι το πρόβλημα στον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό δεν είναι τόσο η συμμετοχή των εργαζομένων και η συναπόφαση. Ε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε 27 ε, διαφορετικά μοντέλα. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι το πρόβλημα της συναπόφασης. Και στις συμβιβαστικές τροπολογίες και σε ολόκληρη την έκθεση τελικά προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια πολύ επικοδομητική προσέγγιση και νομίζω ότι είναι γόνιμη αυτή η συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σογκόρ, θέλετε να πάρετε το λόγο. δεν σημαίνει ότι, το ότι δίνω, δείχνω πράσινη κάρτα δεν σημαίνει ότι ανήκω στους πράσινους. Δεν σημαίνει ότι είμαι με τους πρασίνους, αλλά σε πολλές ε, περιπτώσεις βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα. Για μία ακόμα φορά θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Γκίγκλ, ότι συνεργαστήκαμε καλά και ότι μπορούμε να δεχτούμε όλες τις ε, τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες. Για μας τους Ευρωπαίους είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και λυπάμαι που πρόκειται για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Συμβιβαστήκαμε ε, πολύ τον τελευταίο αιώνα. Συμβιβάσαμε, ε, θέσαμε σε... Κάναμε πολλούς συμβιβασμούς σε σχέση με τις συνεταιρισμούς και ελπίζουμε ότι θα ανανεώσουμε την, ε, το ενδιαφέρον και θα υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους συνεταιρισμούς. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής, θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Εάν βέβαια έχετε υπόψη στις συμβαβιστικές ε, τροπολογίες, εντάξει, θα ακολουθήσετε το δρόμο που ανοίγει το Κοινοβούλιο. Θα... Ε, όποιος δεν μιλάει σημαίνει συμφωνεί. <laughs> Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλες μας οι προτάσεις θα γίνουν στο ακέραιο δεκτές από την Κομισιόν. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση από αυτού. Να ξεκινήσουμε μία συζήτηση μεταξύ των συντονιστών. Θα μου άρεσε ακριβώς επειδή υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ του κλάδου αυτού, να οργανώσαμε μία επαφή με την Κομισιόν για το πώς να προχωρήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα αυτής της έκθεσης, αφού βέβαια την ψηφίσει Ολομέλεια. Χρειάζεται να δώσουμε μια συνέχεια. Όπως είπατε και εσείς, πρόκειται μόνο για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα εναλλακτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να της δώσουμε σημασία, να αυξήσουμε τη σημασία της. Θεωρώ ότι θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι σκιώδεις ε, εισηγητές για να γίνει κάτι τέτοιο. Η ψηφοφορία θα γίνει στο Κοινοβούλιο. και η εργασία αυτή ολοκληρώνει τις εργασίες που έχετε ξεκινήσει για το θέμα της ε, εταιρείας ε, των ε, mutual, των ασφαλιστικών ε, ταμείων. Καμιά φορά όλα αυτά τα θέματα περνούν από όλους και τα προβλήματα εμφανίζονται σε επίπεδο Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε πιστεύω να κλείσουμε αυτό το θέμα και να υπενθυμίσουμε ότι οι συμβιβαστικέ τροπολογίες θα ε, ψηφιστούν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που θα γίνει αύριο. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης για το θέμα των συνθήκων εισόδου των αποσπασμένων εργαζομένων. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Ιακονσάρη. Αναβάλλεται η ψηφοφορία η οποία θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου, αν δεν έχετε αντίρρηση. Επειδή ε, ε, ε, εννοείται φυσικά ότι θα έχει εγκρίνει σήμερα το απόγευμα η Νομική Επιτροπή τη χρονομοδότησή της για την ε, με βάση αυτό το οποίο ζήτησε η δική μας Επιτροπή. Η συγγήτρια θα μπορέσει να σχολιάσει την ε, απόφαση αυτή, η οποία συμπληρώνει τα στοιχεία που συζητήθηκαν στα πλαίσια των συμβαστικών τροπολογιών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήδη ακούσαμε αυτή την γνώμη, τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Θέλω να πω δύο λόγια και μετά να θέσω κάποια ερωτήματα προς την Επιτροπή. Προχωρήσαμε με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Το πρόβλημα ήταν το θέμα της οικοδομής συνειδητοποιούμε ότι στην Ευρώπη, στον τομέα της οικοδομής, των κατασκευών υπάρχει χάος, υπάρχουν δυσκολίες. Άκουσα τις προσδοκίες των εργαζομένων και των εργοδοτών. Ομόφωνα προτάθηκε ο τομέας ε, των κατασκευών να αποκλειστεί από την οδηγία αυτή. Εμείς δεν έχουμε λοιπόν σχετικό, σχετική πρόταση συμβιβασμού γιατί είναι ε, σωστά αιτιολογημένη αυτή η αρχή ότι κανένας τομέας δεν πρέπει μονομερός να αποκλείεται από μια οδηγία. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη θέση αυτή αυτό το οποίο είναι θετικό είναι ότι από φιλοσοφική πλευρά σκοπιά ε, έχουμε μια πολύ σημαντική κατευθυντήρια γραμμή σε αυτή την οδηγία. Υπάρχει ευρία ομοφωνία επί των αρχών και οι διαπραγματεύσεις για τους συμβιβασμούς έχουν προχωρήσει υπό την έννοια ότι όλοι συμφωνούν ότι είναι σημαντική η συμμεταχείριση. Όμως το ερώτημα που, το, που τίθεται είναι πώς θα επιτευχθεί αυτή. Γιατί υπάρχουν και νομικά αλλά και πολιτικά ζητήματα που εκκρεμούν όπως... Τι θα έχει συμβεί με την κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης. Οι διμερείς ε, συμφωνίες είναι ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσει κανείς σε αυτό το τομέα ή μήπως χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ή η εισφορές ε, στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Είναι ένα άλλος δύσκολο τομέα. Χρειαζόμαστε και εδώ ερμηνεία από την Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την άποψη τους επ' αυτού. Σε σχέση με, δηλαδή, τι, θα είναι, τι είναι προτιμότερο, ένας ευρωπαϊκός κανονισμός ή διμερείς συμφωνίες. Ε, που, Πού βρίσκεται η προτεραιότητα από τη σκοπιά του κράτους μέλους, τι θα κάνουμε, θα προχωρήσουμε για προς τη κατεύθυνση της Δημερού συμφωνίας ή προς την ε, ευρωπαϊκή προσέγγιση. Έχουμε ένα ενιαίο κείμενο και εδώ σε αυτό υπάρχει αυτό το βασικό θεμελιώδες ερώτημα το οποίο θα ήθελα να απαντηθεί. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι ορισμοί όπως managers, specialists ή διευθυντές οι ειδικοί. Εδώ έχουμε συμφωνήσει, αλλά εκπαιδευόμενος, τρεινή, εκεί δεν τα έχουμε βρει απολύτως. Υπάρχει μια συμφωνία προς το παρόν τουλάχιστον ανάμεσα σε αυτούς που διαπραγματεύονται. Έχει, έχει γίνει πρόοδος. Το μόνο που μένει είναι οι λεπτομέρειες. Αυτό που βασικά λέμε είναι ναι στην οδηγία, η οποία εντάσσεται καλά στη στρατηγική του 2020. Θέλουμε η Ευρώπη να γίνει μια οικονομία που να βασίζεται στις δεξιότητες, να είναι ένας χώρος ελκυστικός για μορφωμένους, ε, για μορφωμένα στελέχη και ένας χώρος όπου θέλουν οι άνθρωποι με δεξιότητες να εργαστούν. Θέλω όμως να απαντήσω σε αυτές τις βασικές ερωτήσεις Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευτυχώ ακούγονται και φινλανδικά σε αυτή τη συνεδρίαση. Η Λίθα Γιακονσάρη κατέληξε την παρουσίασή τη λέγοντα ότι ο σκοπό τη οδηγία αυτή είναι να ενισχύσει την καινοτομία στην νέα αγορά και οι επιχειρήσεις θέλουν λιγότερη γραφειοκρατία, διότι οι επιχειρήσεις ε, θέλουν να καταστούν δυνατές οι ενδοεπιχειρησιακές ε, μεταθέσεις, ιδίω όταν μιλάμε για αποσπάσει ε, διοικητικών στελεχών και εκπαιδευομένων. Έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά. Διαμορφώσαμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες με θετικό πνεύμα, αλλά δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες μας, γιατί περιμένουμε τη νομική βάση. Μάλλον θα αλλάξει η νομική βάση. Περιμένουμε όμως επιβεβαίωση. Για την οδηγία σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, το βασικό ζήτημα ήταν η σχέση της με τις άλλες βασικές οδηγίες όμως από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η θέση της δικής μου ομάδας. Όπως είπε η Λίσα Γιακονσάρη, δεν υπάρχουν βασικές διαφορές όσον αφορά τους ορισμούς. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Η προβληματική τομή είναι αυτή που ανέφερε η Λίσα και στο ΕΛΚ Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κάποιο συγκεκριμένο τομέα από την οδηγία. Ε, γιατί αν αποκλείσουμε κάποιο τομέα, αυτό μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο και να υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Πάντως, είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε το θέμα όσον αφορά την επικουρικότητα και ίσως αυτό μας επιτρέψει να βρούμε και την κατάλληλη διατύπωση. Η συμμεταχείριση όσον αφορά τους όρους απασχόλησης. Εδώ φαίνεται να προκύπτει μια ξεκάθαρη γραμμή. Για άλλα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και για διμερείς συμφωνίες και για τον κανονισμό 883 για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που ακόμη είναι ανοιχτά. Αλλά ε, μέσα στο γενικότερο πνεύμα συνεργασίας νομίζω ότι μέχρι το Δεκέμβριο το αργότερο θα έχει προχωρήσει αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω σαν συμπλήρωμα αυτά, αυτών που είπε η συγγήτριά μας ότι αν θυμόσαστε οι συντονιστές Ήθελα να, ε, να πάμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για να εξακριβώσουμε τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η πρόταση και ούτως ή άλλως η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επιβεβαίωσε ε, την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημά μας. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Je propose de, de να πάρω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί πάνω σε αυτό το θέμα και για τα θέματα τα οποία θίξατε. Στην πρόταση την οποία υποβάλαμε προβλέψαμε ένα καθεστώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως αφήνουμε μια ευελιξία να συναυτούν διμερείς συμφωνίες. Άρα, επί του παρόντος, μπορεί να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες που να επιτρέπουν οι περιπτώσεις σε περίπτωση ενδοεπιχειρησιακής απόσπασης να υπόκεινται οι εργαζόμενοι στο ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας προέλευσης. Ο κατασκευαστικός τομέας τώρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας και με τις ε, ρυθμίσεις ε, ε, που προβλέπονται, νομίζω ότι μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Τώρα όσον αφορά την ε, ισότητα ευκαιριών, η Κομισιό δεν ήθελε να ευνοήσει οποιαδήποτε ομάδα εργαζομένων, είτε είναι ενδοεπιχειρησιακή απόσπαση, είτε άλλη μεταφορά. Ε, ίσως τώρα όσον αφορά την, την διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών θα έπρεπε να αλλάξουμε κάπως την διατύπωση. Και σας ε, παραπέμπω και στην οδηγία για την ενιαία άδεια που συντάσσεται αυτή τη στιγμή. Και, και έχει οδηγηθεί μια πιο γενική διατύπωση. Τώρα βέβαια η Κομισιό παραμένει στην αρχική της ε, διατύπωση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Η κυρία εισηγήτρια, θα, κυρία εισηγήτρια μάλλον σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση ή όχι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Γιατί θα πρέπει η, η Ευρωπαϊκή Οδηγία να παρουσιάσει μια λογική σε όλα τα κείμενα Δεν θα πρέπει να έχουμε ορισμούς διαφορετικούς σε διαφορετικά κείμενα. Και ούτως ή άλλως έχουμε ήδη οθετήσει αυτή την ενιαία άδεια, το single permit. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Ε, ίσως θα πρέπει να εμπνευστούμε από το πνεύμα του κειμένου για να μην υπάρχουν ε, πολλές προσαρμογές και πολλές ε, ε, εκδοχές του κειμένου. Τι είναι πιο σημαντικό, να δώσουμε προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή στις διμερείς συμφωνίες, διότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Η Κομισιόν θα ήθελε ίσως να ξαναπάρει το λόγο. Όχι. Άρα επί του παρόντος καταγράφεται τις παρατηρήσεις της εισηγήτριάς μας που θα αντικατοπτριστούν και στην γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε στις 5 Δεκεμβρίου. Τώρα στο σημείο 6, για το σημείο 6 δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κοφεράτη, για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση. Παράλληλο θέμα με αυτό το οποίο μόλις συζητήσαμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία, ε, όλους κυρίως τους σκιώδης ηγητές εννοώ, γιατί το θέμα το οποίο μας απασχόλησε είναι περίπλοκο. Και χρησιμοποιήσαμε και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και με τους κοιόδης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Κάτι που μας ε, καθυστέρησε λιγάκι μεν, αλλά που μας επέτρεψε να έχουμε ε, καλύτερα αποτελέσματα, με τα οποία ήταν περισσότεροι σύμφωνοι. Και αυτό είναι καλύτερο από ότι αν προχωρούσαμε μόνοι μας. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε καλύπτουν όλο το, όλο το υλικό, αν όλο το θέμα της οδηγίας και είναι λύσεις που μας επιτρέπουν να πούμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια ρύθμιση που να αποτρέπει την εκμετάλλευση της εποχιακής απασχόλησης ή να, να, να αποτρέψουμε την στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσω της εποχιακής απασχόλησης, διότι και αυτός είναι ο στόχος της οδηγίας. Και ο στόχος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, που αντικειμενικά είναι ευάλωτοι διότι φεύγουν μακριά από τη χώρα τους για να δουλέψουν και από την άλλη πλευρά να αποτρέψουμε η σχέση η επαγγελματική η σχέση, η σχέση εργασίας που δημιουργείται να χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις ε, για, για να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Επομένως, έχουμε προϋποθέσεις που αναφέρονται καταρχάς στον εντοπισμό των διαφορών τομέων, στη διάρκεια ε, του συμβολέου, στις ε, διαδικασίες για να εγγυηθούμε στα άτομα αυτά ε, ένα σπίτι αξιοπρεπές και μετά ο πυρήνας που είναι οι ίσες ευκαιρίες, οι ίσες προϋποθέσεις σε σχέση με τους εργαζομένους των, του κράτους μέλους, των κρατών μελών και να έχουν, να έχουν τους ίδιους μισθούς και κοινωνικές και οικονομικές παροχές αλλά και τις την κοινωνική προστασία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κομμάτι που αφορά τους ελέγχους και τις κυρώσεις. Όταν μιλάω για έλεγχο, μιλάω και για την, την επαλήθευση του σεβασμού των ε, διατάξεων και από την άλλη πλευρά να δημιουργείται και ένας αποθαρρυντικός ε, τρόπο, λόγος ας πούμε. Ε, ούτως ή άλλως θα πρέπει τέτοιου είδους ε, διατάξεις να συνοδεύονται και από ε, προβλέψεις και από διατάξεις να προβλέπουν κάποιες κυρώσεις έτσι ώστε να μην δημιουργούνται οι συνθήκες που θα οδηγούσαν στη μη εφαρμογή της νομοθεσίας, άρα στην μαύρη απασχόληση. Εδώ στον, στον τομέα των εποχια, της εποχιακής απασχόλησης η, η παράνομη εργασία είναι, αποτελεί παράδοση. Και οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές ε, συμφωνούσαν με τις ε, με την οδηγία. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, τα οποία όμως πιστεύω ότι θα λυθούν με τη συζήτηση που θα έχουμε ε, με το Συμβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς δεν ανησυχώ για κάποιες μικρές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, γιατί υπάρχει χρόνος για να τις διορθώσουμε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που σχετικά με το πεδίο εφαρμογής. Γιατί η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χρόνων. Επομένως, δεν αφορά την εποχιακή απασχόληση. Όμως, η οδηγία για την εποχιακή απασχόληση αποκλεί ρητά την δυνατότητα οι διατάξεις ε, να αφορούν τους αποσπασμένους. Υπάρχει μία αντίφαση, για την οποία δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι, αλλά υπάρχει στις οδηγίες. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να την επιλύσουμε, ε, καταλήγοντας σε μία συμβιβαστική τροπολογία που θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική θέση με το Συμβούλιο, έτσι ώστε να επιλύσουμε αυτή την αρχική αντίφαση που υπήρχε. Εγώ πιστεύω ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταλήξουμε σε μία λύση ε, στα πλαίσια της αυριανής ψηφοφορίας, έτσι ώστε να έχουμε τροπολογίες με τις οποίες όλοι να συμφωνούμε και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα γίνουν ε, όταν ε, συζητήσουμε το θέμα με το Συμβούλιο έτσι ώστε όταν ολοκληρωθεί αυτή όλη αυτή η διαδικασία να έχουμε μία σειρά διατάξεων σαφέστατες να μην χρειάζεται να ερμηνεύσουμε τις διατάξεις διότι η ερμηνεία της διάταξης οδηγεί στην μη πιστή εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί και καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι ένας, ε, ένας φιλόδοξος στόχος, η δουλειά δεν είναι εύκολη, αλλά αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, εάν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ε, τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας, νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και να προσπαθήσω να σας δώσω περαιτέρω τελικές διευκρινήσεις για κάποια σημεία πάνω στα οποία έχουμε καταλήξει σε ευρύτερες συμφωνίες, συμβαστικές ε, συμφωνίες. Προσπαθήσαμε μέχρι και τελευταία στιγμή να, βρούμε, να, να πετύχουμε μια συμφωνία και ε, η συμφωνία αυτή οφείλεται στο πάθος και στο ενδιαφέρον που έδειξαν όλοι και οι σκιώδη και άλλοι συνάδελφοι διότι μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει τον κόπο και για την προσοχή και την προσοχή και την, ε, τον κόπο που κατέβαλαν οι συνάδελφοι. Κυρία Τουρίνεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν πολύ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε στην έκθεση αυτή. συμφωνούμε και είμαστε ικανοποιημένοι εμείς ως πράσινοι με την δουλειά αυτή. Την προηγούμενη συνεδρία, αν δεν απατώμε, συμφωνήσαμε επί ενός πακέτου. Μέσα εκεί σαφώς υπάρχουν πράγματα που σου αρέσουν και άλλα που σου αρέσουν κάπως λιγότερο. Αυτό είναι φυσιολογικό στις ε, διαπραγματεύσεις. Δίνει κανείς αλλά και παίρνει. Εμείς ε, οι πράσινοι θα θέλαμε μεγαλύτερη βελτίωση, με περισσότερες βελτιώσεις σε αυτή την οδηγία, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που υπάρχει τώρα και πιστεύω ότι όλες οι ομάδες συμφωνούν με τις βασικούς συμβιβασμούς. Τέσσερα είναι τα πολύ σημαντικά θέματα για μας και τα επισημάναμε σε όλη τη διαδικασία. Χαιρόμαστε που ε, περιλήφθησαν πρώτον η αρχή της ίσης μεταχείρισης, την οποία ε, πραγματικά καταφέραμε να επιτευχθεί, να συμπεριληφθεί. Δεύτερον, είναι πολύ καλό το κείμενο αυτό και τα άρθρα για την στέγαση. Τρίτον, για τις κυρώσεις από το κείμενο της Κομισιόν γινόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών. Μας αρέσει αυτό. Έχουμε συμπεριλάβει και τους υπεργολάβους. Και τέταρτον, το θέμα της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων. Το επισημαίνουμε αυτό. Θα θέλαμε να προχωρούμε λίγο περισσότερο, δηλαδή ένα ε, ποσοστό 20% ο αριθμός που συμπεριλήφθη είναι χαμηλότερος, αλλά χαιρόμαστε που Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα τμήμα που αφορά την παρακολούθηση της στήρησης. Εάν δεν φροντίζουμε για την εφαρμογή και την παρακολούθηση τη της στήρησης της νομοθεσίας, ε, ε, η νομοθεσία αυτή χάνει από την αξία της. Χαιρόμαστε λοιπόν ότι που μπορούμε να συμφωνήσουμε με ε, αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπαλτασάρη και μετά κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει εξαιρετική εργασία. Κυρίως ε, για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι είχαμε δύο αντιφατικά θέματα τα οποία έπρεπε να συμφιλιώσουμε. Το, ίδιο, το ένα ήταν ότι έπρεπε να, υπερασπίσουμε κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι αντικειμενικά αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης, δεν τους πληρώνουν αρκετά χρήματα και ε, εργάζονται και ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες και από την άλλη πλευρά η, η εποχιακή απασχόληση ε, πρέπει να ρυθμιστεί, πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνει όποια, όλες, ε, όλες τις κοινωνικές καλύψεις, ε, ό,τι προβλέπει το κράτος δικαίου, το κράτος πρόνοιας, ε, το συγκεκριμένο. Δηλαδή θα έπρεπε ό,τι προσφέρει το κράτος πρόνοιας στους υπηκόους του να το προσφέρει και στους εποχιακούς εργαζομένους. Άρα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη δουλειά με τους σταφείς, με σαφείς στόχους. Πετύχαμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες με τις οποίες όλοι είμαστε σύμφωνοι και στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων λύσαμε και ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπήρχε μια σύγχυση ανάμεσα στον αποσπασμένο εργαζόμενο και στον εποχιακό εργαζόμενο. Είναι ε, ζωτική σημασία, ήταν ζωτική σημασία να διευκρινίσουμε τους όρους, να ξέρουμε δηλαδή σε τι αναφέρεται η νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά τώρα παραμένουν όμως δύο απορίες. Η μία είναι η συμβαστική πρόταση G, για την μετα... δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και την κοινωνική κάλυψη που συμπίπτει με την διαμονή. Αυτό είναι μια, μια αρχή η οποία είναι επιβεβαιωμένη. Όταν γίνεται η μεταφορά δηλαδή με βάση όλες, όλες τις ε, ε, διαδρομές που ακολουθεί ο, ο εποχιακός εργαζόμενος. Ε, εκεί μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνο, κίνδυνος να δημιουργηθεί μια κάποια σύγχυση, δηλαδή να, επιδι, να επιβαρυνθεί ε, το κράτος μέλος υποδοχής με κάποιους μηχανισμούς ε, τους οποίους ούτως ή δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει και μετά η συμβαστική τροπολογία B όπου, όπου η λέξη may δεν μας καλύπτει διότι μιλάμε για τον, για τον εργοδότη και τον υπεργολάβο υπάρχει ο, εργοδό, εργοδότης και ο εργοδότης δεν μπορεί να ε, ταυτίζεται αυτόματα με τον υπεργολάβο γιατί υπάρχει και μία οδηγία ούτως ή άλλως το 2000 όπου ε, προβλέπονται πολύ συγκεκριμένα οι διακριτή ρόλοι του εργοδότη και του υπεργολάβου. Έχουν διαφορετικές ε, υποχρεώσεις ο ένας και ο άλλος. Επομένως θα πρέπει αυτά τα θέματα ευθύνη του ενό και του άλλου να τα διευκρινίσουμε, διότι δεν είναι λογικό ένας εργοδότης ο οποίο δεν γνωρίζει τι κάνουν οι υπεργολάβοι του να πρέπει να πληρώσει ο ίδιο. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω και ελπίζω να μπορέσουν να, να τα διευκρινίσουμε μέχρι αύριο. Κατά τα λοιπά, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έχουν γίνει και μπορούμε να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να ε, διευκρινιστούν αυτά τα δύο και τα δύο ζητήματα τα οποία παραμένουν σε κρεμότητα. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά η κυρία Μάρκη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ ικανοποιητική εργασία που έχει γίνει και σε πολλές βασικές τροπολογίες εκτιμούμε ότι στο τέλος μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι κοινό. Υπάρχουν πολλές καλέ συμβασικέ τροπολογίε. Ε, και νομίζω ότι τον έφερε ο συνάδελφο Μπαλτασάρη ότι πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των εποχικά εργαζομένων αφενό και των αποσπασμένων αφετέρου. Συχνά ε, αναφερόμαστε σε αυτά από κοινού και πρέπει σαφώς ε, να τα διαχωρίσουμε. Και θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα, κύριε Κοφεράτη με την ε, τροπολογία μου 106 τι έχει γίνει. Υπάρχει σε κάποια συμβιβαστική τροπολογία. Εκεί επισήμανα ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την δυνατότητα ε, να αρνούνται αιτήσει ε, εάν δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στη συγκεκριμένη χώρα για παρόμοιους ε, εργαζόμενους τη χώρα. Την τροπολογία μου 106 δεν την έχω βρει κάπου, εκτός αν στις διαπραγματεύσεις μετατοπίστηκε κάπου αλλού, σε κάποια άλλη συμβαστική τροπολογία. Θα με ενδιαφέρε μια απάντηση από αυτού. Με τις τροπολογίε δεν έχω εγώ ιδιαίτερα πρόβλημα. Ανέφερε την Τζέι ο συνάδελφο ε, Μπαλκασάρε νομίζω ότι μέχρι την ψηφοφορία θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια άκρη. Μόνο στην τροπολογία, επαναλαμβάνω, 106 έκαναν καλές προτάσεις οι συνάδελφοι για τις υπόλοιπες τροπολογίες. Μόνο για την 106 θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ε, Πρόεδρος, προτείνω να σας απαντήσει στο τέλος ο εισηγητής όταν θα απαντήσει και στα υπόλοιπα σχόλια. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ε, όλο το προσωπικό για τις ε, ειλικρινείς προσπάθειες που κατέβαλαν να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες γιατί δεν ήταν εύκολο αλλά νομίζω ότι καλά τα καταφέραμε. Παραμένουν ένα-δύο μικρά σημεία στη συμβαστική τροπολογία Α και στην J, γιατί περί του ιδίου θέματος πρόκειται και στις δύο αυτές τροπολογίες. Πάλι επανερχόμαστε στο θέμα των εργαζομένων, του αν υπάρχονται στην οδηγία για την απόσπαση ή στην οδηγία για τους εποχικά εργαζομένους. Νομίζω ότι εδώ το θέμα έχει σχέση με το ότι οι εποχικά εργαζόμενοι μπορούν να αποσπώνται, αλλά εάν αποσπώνται ε, ε, υπάγονται στην οδηγία για τους αποσπασμένους. Και στην τελική πρόταση, στη συμβιβαστική τροπολογία Α και J, πρέπει να δούμε πώς θα την τροποποιήσουμε, γιατί δεν μας διευκρινίζει την κατάσταση. Θα μπορούσε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η δική τους θέση. Νομίζετε ότι αυτή η τελευταία πρόταση διευκρινίζει την κατάσταση. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατάσταση. Δεν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το οποίο τώρα έχουμε μας προσφέρει την ξεκάθαρη κατάσταση που θα επιθυμούσαμε. Για την τροπολογία F, για την ίση μεταχείριση, μπορούμε να την υποστηρίξουμε και την τροπολογία G. Και έχω άλλα δύο σχόλια για την συμβαστική τροπολογία S, για το άρθρο 16 που είναι και ο πυρήνα αυτού του νομοθετήματο. Στο τρίτο τμήμα, για τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 883 του 2004, ζητήσαμε από τον εισηγητή να μπει η εξή φράση. Όταν βασίζεται στην δραστηριότητα απασχόλησης του εποχικά εργαζομένου. Αν δεν γίνει αποδεκτό αυτό, πιστεύουμε ότι κάπως η δραστηριότητα ε, του εποχικά εργαζομένου κάπως πρέπει να συνδεθεί με, τα, με τις παροχές κοινωνικής ασφαλείας. Καταλαβαίνουμε τα υπόλοιπα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο. Και τέλος, για την συμβαστική τροπολογία H, υποστηρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εθνική νομοθεσία θα δίνει επαρκείς πόρους ε, τις αρχές που θα διεξάγουν ελέγχους και επιθεωρήσεις και πρέπει να έχουν και το κατάλληλο προσωπικό. Όμως, μια φράση που λέει ότι επίσης τα αποτελέσματα των προηγούμενων επιθεωρήσεων συλλέγονται και είναι αντικείμενο επεξεργασίας για την σωστή εφαρμογή της οδηγίας είναι μια φράση κάπως υπερβολική πιστεύω. Δεν λέω ότι ξεπερνάει το όριο για μας, ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή του αποδεκτού, αλλά θα ήταν προτιμότερο να δούμε, ε, αν μπορούμε να πούμε, αν υπάρχουν επαρκείς πόροι και προσόντα. Ε, αυτό αρκεί για να πληρούν τα κράτη-μέλη τις ε, υποχρεώσεις τους. Όπως σας είπα όμως, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της Επιτροπής για την τελευταία πρόταση της συμβαστικής τροπολογίας Α και J. Πιστεύει η Επιτροπή ότι διευκρινίζεται η κατάσταση με αυτό ή όχι. Και άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη για τις ε, ειλικρινείς του προσπάθειες να καταλήξουμε σε συμφωνία για την έκθεση αυτή. Ο κύριος Μπεναβιάς και μετά η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτό είναι το είδος της έκθεσης οδηγίας που δίνει την εικόνα στους συμπολίτες μας ότι σε κάτι είμαστε κι εμείς χρήσιμοι. Ε, και τώρα αυτό το οποίο κάνουμε το χρήσιμο πρέπει κανείς να προσπαθεί να αποφύγει το τέλειο αν θέλει να πετύχει κάτι το καλό λοιπόν να μην ε, σπάει κανείς το κεφάλι του τι είναι ε, ο αποσπασμένος σε σχέση με τον εποχιακό. Εν πάση περιπτώσει μπορεί κανείς να είναι και αποσπασμένος και εποχικός και το αντίστροφο. Εν πάση περιπτώσει θέλω να συγχαρώ και τον εισηγητή και όλους όσοι κατέληξαν στους συμβιβασμούς και θα υπερψηφίσω την έκθεση. Η, η Ένωση εν μέσα στις διαφορετικές απόψεις, λέει η Πρόεδρο. Γιαζοβγισκά είναι το όνομά σας, κυρία. έκανα λάθος το όνομά σας, γιατί ξεκινάει από «για». Από «για». Εντάξει, εντάξει. Κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι το όνομά μου είναι πολύ δύσκολο γεια απο γεια. ενταξει ενταξει κυρια προεδρε ξερω οτι το ονομα μου ειναι πολυ δυσκολο για ορισμενους ε, Δεν, δεν με ενοχλεί. Δεν πειράζει. Μπορώ επιτέλους να πω και εγώ την άποψή μου. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που έχουν επιφυλάξεις για τη συμβιβαστική πρόταση J. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα αποκλειστούν από το Συμβούλιο από ό,τι μοιάζει. Και όσον αφορά την τροπολογία G, το ε, τελευταίο μέρος που αφορά την ε, ε, επιστροφή, την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να πούμε ότι σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σε, αυτού, σε, σε τέτοιους καιρούς κρίσης δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να προσθέτουμε τέτοιου είδους διατυπώσεις. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Έκλεισε λοιπόν, ε, εξαντλήθηκε ο κατάλογος των ομιλητών που είχαν ζητήσει αυτό που είχαν ζητήσει το λόγο. Θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω απλώς να απαντήσω σε ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν σε σχέση με την ορική σκέψη 9 στο άρθρο 2.2 που γίνεται αναφορά την ε, οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων αλλά και την ε, οδηγία για τους εποχικούς και την ειδική άδεια. Πράγματι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης γιατί οι αποσπασμένοι ε, αναφέρονται σε αυτήν την οδηγία και όταν μιλάει κανείς απόσπαση από το ένα κράτος μέλος σε άλλο ισχύει αυτή η οδηγία. Μην ξεχνάμε ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι στους οποίους αναφέρεται η οδηγία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν άμεση σύμβαση με τον εργοδότη τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Σιγητής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους κοιόδης συζητητές για τις παρατηρήσεις που, ήθελαν, που θέλησαν να κάνουν. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και έχουμε λίγο χρόνο στο, διάθεσή μας για να βρούμε τις τελευταίες ε, τροποποίησεις ε, στην διατύπωση για να συμφωνήσουμε όλοι. Θα ήθελα τώρα, να, εν συντομία, να ασχοληθώ με κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Η πρώτη ερώτηση για το πεδίο εφαρμογής. Μπορούμε να καθορίσουμε το κείμενο ε, μέσω των σκιωδών εισηγητών. Όμως, παρόλα αυτά, το πρόβλημα υπέ, υπάρχει, διότι οφείλεται στο τρόπο με τον οποίο είναι συνταγμένε, είναι διατυπωμένε οι δύο οδηγίε. Ένα λέγεται ότι ένας αποσπασμένος εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι εποχιακό. Και αυτό το συμφωνώ κι εγώ, αλλά αυτή δεν είναι η άποψή μου. Δεν έχει, συγγνώμη, δεν έχει καμία σημασία η άποψή μου. Αυτό που μετράει είναι το κείμενο των οδηγιών. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, έχουμε μία διατύπωση που να λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα εργαζόμενο ο οποίος να καλύπτεται από τις δύο οδηγίες ή να υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος να μην καλύπτεται από καμία από τις δύο. Μιλάμε για μικρό αριθμό ε, ενδιαφερομένων βέβαια, αλλά όταν πρόκειται για ένα δικαίωμα είτε οι ενδιαφερόμενοι είναι 10, είτε είναι ένα εκατομμύριο, κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλουμε είναι σημαντική, αλλά μπορούμε να την καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Δηλαδή να έχουμε μία διατύπωση που θα μας επιτρέψει στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε μετά με το, με το Συμβούλιο να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να λύσει οριστικά αυτό το μικρό συμβάν το οποίο εμφανίζεται στην διατύπωση των δύο οδηγιών. Τώρα, όσον αφορά μια άλλη παρα... τις άλλες παρατηρήσεις που έγιναν, παραδείγματος χάρη, Συμβαστική τροπολογία G. Το κείμενο είναι μεγάλο εδώ σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία και θα πρέπει να βρούμε και όταν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε συνθετικά ένα, ένα επιχείρημα κάπως μπερδευόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι ο πυρήνας της συμβαστικής πρότασης G, πάνω στον οποίο συμφωνήσαμε από την αρχή όλοι, είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν δικαιώματα αναγνωρισμένα και απαιτητά που να είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τους εποχιακούς εργαζόμενους του κράτους μέλους. Δεν θα πρέπει βέβαια να αποδυναμώνεται η πολιτική άποψη των μεν και των δε. Και εάν μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμα περαιτέρω το κείμενο, ευχαρίστως. Εάν τον, τα, τα, τα, τα συμπυκνώσουμε πάρα πολύ τα πράγματα, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Π.χ. αυτό που είπε ο συνάδελφος Μπαλταζάρ για την συμβιβαστική πρόταση P που αφορά τις ευθύνες τις διαφορετικές συνθήκες, υποχρεώσεις ανάμεσα στον εργοδότη και στον ε, υπεργολάβο. Η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σωστή και, την, ε, και, και με βρίσκει σύμφωνο, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι στη σύνθεση που γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας ε, βοηθούν οι διαφορετικές γλώσσες. Αυτό το οποίο είναι κατανοητό στα Ιταλικά και αυτό είναι εκπληκτικό βέβαια, διότι τα Ιταλικά δεν είναι μια γλώσσα που επιτρέπει να διατυπώνουμε ε, συμπυκνωμένα, αν θέλετε, ε, κάποιο πράγμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται σαφές στα Ιταλικά δημιουργεί προβλήματα στα Αγγλικά. Βέβαια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διατύπωση με την οποία να συμφωνούν όλοι. Αλλά τέλος πάντων είναι πιθανόν να υπάρχει διαφορετική υποχρέωση για τον εργοδότη και τον ενδεχόμενο υπεργολάβο. Διότι ο τελευταίος στην αλυσίδα μπορεί να διαπράξει ένα αδίκημα, μπορεί να μην εφαρμόσει την ε, διάταξη, καλόπιστα βέβαια, διότι μπορεί να μην τον έχει ενημερώσει ο εργοδότης ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία ή μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Επομένως δεν μπορούμε να, θεωρήσουμε, θεωρήσουμε αυτόματα υπεύθυνο χωρίς να διευκρινίσουμε αυτή την διαφορά. είναι λογικό ο καθένας να πληρώνει, αν θέλετε, για τις ευθύνες που αναλαμβάνει. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση, μία διόρθωση που να αντικατοπτρίζει τη συμφωνία των σκιωδών εισηγητών. Ίσως ο Μπαλταζάρ και εγώ, επειδή μιλάμε και οι δύο, είμαστε και οι δύο Ιταλοί, ε, καταλήξαμε σε μια απλούστευση η οποία ενδεχόμενα να μην ε, έγινε κατανοητή από τους άλλους συναδέλφους. Εκεί χάσαμε λίγο στα χαρτιά. Θα το βρούμε όμως. Τώρα, το 106 θεωρήθηκε απαράδεκτο και στο κείμενο θα το δείτε. Θα δείτε και για, για ποιους λόγους ε, η τροπολογία αυτή δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Α, μία τελευταία παρατήρηση όπως είπε και η συνάδελφος το Ρούνεν, αλλά και το αναγνώρισαν και οι άλλοι συνάδελφοι, καταβάλαμε μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν θα ήθελα, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ε, να, δούμε στο στο τέλος ποια είναι η διάταξη την οποία θα πρέπει να προσαρμόσουμε και να διορθώσουμε για να πετύχουμε συμφωνία και να ξεχάσουμε τα όσα έχουμε κάνει πιο πριν. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε συμφωνία και πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθη λόγω του ότι ήταν όλοι διαθέσιμοι, ότι όλοι έδειξαν θέληση να βρεθεί μια ε, συμφωνία και ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο μπορεί να γίνει. Αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι να ε, μπορούμε να βρούμε μια λύση για ένα πολύ σημαντικό θέμα κατά την άποψή μου και θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Κομισιό από θέση ισχύω κατά την άποψή μου διότι δεν μπορεί να αγνοήσει την, τις απόψεις μας έτσι όπως θα διαμορφωθούν αύριο και κυρίως όταν και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφασίσει και όταν περάσει από την Ολομέλεια. Πάντως εγώ πιστεύω ότι ναι μεν μπορεί να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω αλλά αυτό το οποίο έχουμε, στο οποίο έχουμε καταλήξει τώρα είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι αύριο πρέπει να κάνουμε κάποια μικρή προσαρμογή και αν μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε και τις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Εν πάση περιπτώσει θα ψηφίσουμε αύριο. Φτάσαμε λοιπόν στην επιστολή για την ενεργοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και όπως σας έχω ήδη πει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 Πολύ καλά. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη... Ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη επιστολή που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αφορά την Πορτογαλία. στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιοχή Νόρτε Τσέντρο. Στο σχέδιο αυτό επιστολής μας προτείνεται μία πρόταση τροπολογίας την οποία θα θέσω σε ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας αυτή που σκοπό έχει να εισαχθεί μια νέα παράγραφος 8α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Έχετε όλες τις κάρτες σας. Επαλήθευση. Ποιος δεν έχει κάρτα. Δύο σοσιαλιστές είναι κακοί μαθητές. Και Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άλλοι έχετε τις κάρτες σας, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. 36 υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, 21 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Το σύνολο της επιστολής. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Όχι, δεν χρειάζεται. Άρα ψηφίζουμε επί του συνόλου της επιστολής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη δεύτερη επιστολή που αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ η, η, περιοχή είναι το Άλτο Ατίτζε. Δεν υπάρχει τροπολογία στην περίπτωση αυτή. Η ομάδα εργασίας έχει ομόφωνα συντάξει την επιστολή Άρα ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, η δεύτερη αυτή επιστολή εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα υποδεχτούμε τον κύριο Σελ, ο οποίος εκ μέρους της Κομισιόν θα μας παρουσιάσει την σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων συμπεριλαμβανομένου και του FSF. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, σας ζητώ να αρχίσουμε και πάλι τις εργασίες μας, ε, να υποδεχτούμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και να ασχοληθούμε χωριστά, καταρχήν με την νομοθεσία που ονομάζεται οριζόντια νομοθεσία, στο συνολικό πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και κατόπιν να ασχοληθούμε με την ε, νέα πρόταση για την ε, κοινωνική καινοτομία. Έχετε το λόγο για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω καταρχήν να παρουσιάσω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο συνολικό του πλαίσιο. Όπως γνωρίζετε, τον, φέτος τον Οκτώβριο, στις αρχές Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πακέτο των διαρθρωτικών ταμείων που συμπεριλαμβάνει τους κανονισμούς που θα πρέπει να ισχύσουν για το διάστημα 2014 έως 2020. Στην συνολική ανακοίνωσή της, η Κομισιόν ανέφερε ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές αυτής της μεταρρύθμισης. Πρώτον, ότι θα πρέπει να συσχετιστούν με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 με τρόπο συγκεκριμένο. Δεύτερον, ότι πρέπει να δίνουν έμφαση στα αποτελέσματα, να υπάρξει καλύτερο συντονισμό, εναρμόνιση και ε, συνεργασία μεταξύ των διαθέσιμων ταμείων και ότι θα πρέπει να ε, λειτουργούν περισσότερο στον τομέα της εταιρικής σχέσης. Και αυτά όλα θα σας τα εξηγήσω σε λίγο. Καταρχήν λοιπόν υπήρχε αυτή η γενική ανακοίνωση που αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο η οποία είχε ήδη παρουσιαστεί τον Ιούνιο. Μία από τις ε, ως μία από τις εφαρμοστικές προτάσεις ήταν ε, το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων. Το, το νέο στοιχείο εδώ είναι ότι υπάρχει ένας γενικός κανονισμός που καλύπτει και το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και το Ταμείο ε, γεωργικής ανάπτυξης και το Ταμείο ε, της Αλίας. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια πραγματικού συνδυασμού σε έναν κανονισμό όλων των γενικών διατάξεων που ισχύουν στα ταμεία αυτά. Μια προσπάθεια απλούστευσης και εναρμόνισης. Ο Γενικός Κανονισμός περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεις που αφορούν όλα τα ταμεία την ιδέα, ας πούμε, ότι θα πρέπει να προχωρούμε προς μια ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη και έτσι για να πλουστεύσουμε την κατάσταση δεν θα πρέπει κάθε ταμείο να πηγαίνει σε μια χώρα ή σε μια περιοχή και να ξεκινά τις διαπραγματεύσεις εκεί, αλλά να γίνεται συνολική συζήτηση με όλα τα ταμεία για μια ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό ε, καθορίζει τις σχέσεις με τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Ε, εντοπίζει την ανάγκη να, ε, να περιοριστούν οι τομείς προτεραιότητας, να υπάρχει στόχευση. Αυτός ο κανονισμός είναι πολύ πιο... Ε, έχει μεγαλύτερη μορφή καθοδήγησης από ότι οι προηγούμενοι κανονισμοί. Δηλαδή θέλει να πάρει τις περιφέρειες από το χέρι και με τρόπο ε, εταιρικό να καθοδηγήσει την κατάσταση. Στον κανονισμό αυτό υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανονισμοί ανά ταμείο. Ένας από αυτούς αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι ένας αρκετά περιορισμένος κανονισμός, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ουσίας περιλαμβάνεται στον γενικό κανονισμό που αφορά όλα τα ταμεία και μόνο κάποιες συγκεκριμένες παράγραφοι και κάποια άρθρα ε, αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αν δείτε την κάλυψη και θα δείτε μια άλλη καινοτομία. Υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα σε τριών ειδών περιφέρειες. Αυτές που έχουν κατακεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 75%, αυτές που έχουν κατακεφαλήν ΑΕΠ από το 75% έως 90% και οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες που λειτουργούν σε επίπεδο πάνω από το 90% κατακεφαλήν του ΑΕΠ. Ε, αυτό θα έχει σημασία μετέπειτα, όπως θα διαπιστώσετε, ε, από τα, τις απαιτήσει των προγραμμάτων που θεσπίζονται για κάθε είδος περιφέρειας. Αν δείτε τώρα τα ποσά. Για το σύνολο του 2014-2020 για τα διαρθρωτικά ταμεία μιλάμε για ένα ποσό 376 δις. Αυτό είναι το συνολικό ποσό λίγο ε, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υπάρχει ένα ελάχιστο μερίδιο. Αυτό εισάγεται για πρώτη φορά. Διαπιστώσαμε ότι σύν το χρόνο το ποσοστό του ταμείου έχει πέσει από το 40% στο 22%. Αυτή η τάση θα πρέπει να αντιστραφεί. Και γι' αυτό θεσπίσαμε ένα ελάχιστο 25% του συνολικού πακέτου συνοχής, δηλαδή 84 δις. Αυτό στηρίζεται βασικά στο ότι έχουμε μια στρατηγική Ευρώπης 2020, έχουμε τους ε, πρωταρχικούς στόχους όπως να φύγουν 20 εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια ή το 75% τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού να είναι ενεργό στην αγορά εργασίας και αυτή η πρωταρχική, αυτή η βασική στόχη θα πρέπει να στηρίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, πρόκειται σαφώς για ένα ελάχιστο. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. στο 25% τα 84 δις λοιπόν συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσό 2,5 δισεκατομμυρίων που θα καλύψει το διάδοχο του κανονισμού της, των τροφίμων για τους ε, στερημένους, Food for the Deprived, που συζητείται τώρα να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση για την επόμενη διετία. Όμως για μακροπρόθεσμα ε, προτείνεται να συμπεριληφθούν 2,5 δις ε, αυτού του προγράμματος στα 84 δισεκατομμύρια που είναι το 85% του Ταμείου Συνοχής. Αυτά όλα είναι υποσυζήτηση. Δεν ξέρουμε άμεσα στο μέλλον ποιο θα είναι η τύχη αυτού του μέτρου και δεν ξέρουμε και μακροπρόθεσμα τι θα γίνει. Βλέπω ε, ότι κάποιοι από εσά χωρίς να μιλάτε δείχνετε να ξέρετε τι θα συμβεί ή έχετε μια εικόνα του τι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει πρέπει όλα αυτά να επαληθευτούν και από το Συμβούλιο. Αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για να ε, συνδεθούν με την ιδέα μας περί προτεραιοτήτων, έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Ξεκινάμε από ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο προχωράμε σε σύμβαση εταιρική σχέσης και σε ε, επιχειρησιακά προγράμματα. Υπογραμμίζω, εδώ υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των ταμείων. Όλα θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, άρα κατά προτίμηση μία εταιρική σύμβαση. Δεν ξέρω αν οι χώρες θα επιλέξουν μία σύμβαση αναχώρα ή μία ε, σύμβαση ανά ε, περιφέρεια αλλά πάντως αυτός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουμε. Τα επιχειρησιακά προγράμματα θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Αν δείτε τώρα την επόμενη διαφάνεια θα διαπιστώσετε ότι εδώ λαμβάνεται υπόψη η ενίσχυση του ολοκληρωμένου προγραμματισμού. Υπό τις παρούσες συνθήκες έχουμε ε, μια προσέγγιση ενός ταμείου και θέλουμε να υπάρχει να υπάρξει αλλαγή σε σχέση με αυτό που συνέβη στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση αν δεν έχουμε προσέγγιση πολλα, πολλών ταμείων. Αυτό θα επηρεάσει τη δουλειά που θα γίνεται και επιτόπου στις περιφέρειες και τις χώρες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα απαιτηθεί βαθιά συνεργασία ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις και ίσως να επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα συζητηθεί αυτό αργότερα ε, στους κοινοβουλευτικούς χώρους. Τώρα, στο θέμα της ex ante conditionality that is mainly the check της συμμόρφωσης. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει οι περιφέρειες να μπορούν να χειριστούν τα χρήματα. Αν οι προϋποθέσεις ε, δηλαδή ε, βοηθούν την κίνηση, τότε ε, προτείνεται να υπάρξουν μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, με όλους τους παράγοντες που ενσωματώνονται σε αυτήν, ό,τι έχει γίνει για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης έτσι ώστε με τρόπο συντεταγμένο να ε, συμπεριληφθεί στην μακροοικονομική ε, κατάσταση. Αν διαβάσετε τα άρθρα του Six ε, δεν λένε κάτι τέτοιο. Οι, μακροοικονομικ... οι αντιδράσεις ε, της μακροοικονομικής συμμόρφωσης ε, προκαλούνται από μια αλληλουχία γεγονότων. Δεν μπορεί μόνη της η Κομισιόν να, να ενεργοποιήσει αυτές ε, τις ε, διαδικασίες. Στηρίζονται πάντοτε σε απόφαση του Συμβουλίου. Μιλάμε πάντοτε για μια αλληλουχία. Δεν εμφανίζεται με ευνίδιο τρόπο ο τρόπος που, το προτείνεται τώρα ευθυγραμμίζεται και με το six pack. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένας αυστηρότερος τρόπος χρήσης των πόρων, ώστε και η Κομισιόν να αναλαμβάνει την ευθύνη του προγραμματισμού για κάποιο κράτος μέλος υπό ορισμένες συνθήκες ώστε να φροντίσει ότι το, να χρησιμοποιηθούν οι πόροι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις συστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα ε, από που ξεκινούν από την οικονομική διακυβέρνηση. Στο μακροοικονομικό χώρο δίνεται έμφαση στα αποτελέσματα. Λειτουργούμε με βάση ένα πλαίσιο επιτευγμάτων, επιδόσεων και η εικόνα αυτή πρέπει να είναι σωστή. Επ, αυτών συμφωνούμε και με τα κράτη-μέλη και με τις περιφέρειες. Από την ώρα όμως που θα αποφασιστεί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Και αν δεν υπάρχει ε, συνέπεια θα υπάρξουν συνέπειες. Υπάρχουν διακοπές και αναστολές. Όταν μια χώρα ξεφύγει στην καθημερινή οικονομική διαχείριση θα υπάρχουν διακοπές και αναστολές και αυτό διευκολύνει το ότι ε, μέσα στο 2010 έχουμε φτάσει σε ποσοστό σφάλματος κάτω από το περίφημο 2% που μας έχει δώσει μια διαβάθμιση α από το ελεγκτικό συνέδριο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τα προσεγγίζει όλα αυτά μόνο από τη σκοπιά της, της ε, πολιτικής. Πρέπει να λάβει υπόψη και την δημοσιονομική διαχείριση και την κάθε χώρα ξεχωριστά. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αποθέματα επιδόσεων ε, ε, αποθεματικά τα οποία θα πρέπει να ε, αποφασίζονται στο ξεκίνημα του προγράμματος και θα αφορούν κάθε χώρα συγκεκριμένα. Δεν θα μπαίνουν δηλαδή σε κάποιο ε, μεγάλο ευρωπαϊκό απόθεμα και αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επιδόσεων στο δεύτερο ήμιση της προγραμματικής περίοδου. Αυτό που θέλουμε να εισάγουμε είναι μια, την έμφαση στα αποτελέσματα. Θέλουμε να εισάγουμε την δυνατότητα να υπάρχουν εκ των προτέρων καθορισμένα αποτελέσματα, δηλαδή κατάρτιση δασκάλων, εκπαίδευση σε ένα πρόγραμμα 2.000, 2.000 δασκάλων και υπάρχει ροή πόρων εάν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με επιτυχία. Και αυτό συνδυάζεται με κάποιο άλλο θέμα που αποτελεί απλούστευση. Αν μπορέσουμε να καταλήξουμε εκ των προτέρων σε, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση 2.000 ε, δασκάλων και δεν θα αρχίσουμε να ελέγχουμε τα, τις δαπάνες τους για ταξίδια, για μετακίνηση. Δηλαδή θα ελέγχουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Η άλλη προσπάθεια πλούστευσης είναι η εναρμόνιση των κανόνων, τα κοινά σχέδια δράσης και η μείωση του ελεγκτικού άχθους. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την απλούστευση σε κάθε επίπεδο για μας την εναρμόνιση των κανόνων για τη χώρα που επίσης είναι η εναρμόνιση των κανόνων, αλλά και η, το να δουλεύουμε με τελικά αποτελέσματα διευκολύνει και τη δουλειά και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και βεβαίως μειώνει το ελεγκτικό άχθος που και αυτό είναι σε όφελος του τελικού δικαιούχου. Προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε και να ενσωματώσουμε τις απλουστεύσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η εταιρική σχέση στην οποία αναφέρθηκα, η οποία θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση σε κάθε επίπεδο και σε κάθε φάση του προγράμματος. Για να μπορέσει να λειτουργήσει, σκεφτήκαμε να εισάγουμε ένα κώδικα δεοντολογίας, ένα κώδικα συμπεριφοράς για το πώς θα συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε όχι μόνο τα κράτη-μέλη να έχουν ίση μεταχείριση, να δουν πώς θα εφαρμόσουν αυτή την εταιρική ε, σχέση, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να ε, θεσπίσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας για έναν κοινό προγραμματισμό και για την κοινή εφαρμογή. Αυτός ο κώδικας λοιπόν συμπεριφοράς αφορά όλους τους εταίρους. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και αυτό βοηθά στο να δημιουργηθούν δυνατότητες. Ε, έχω δει πολλά άσχημα πράγματα σε ε, τρίτες χώρες ε, για τη, το θέμα της διοίκησης αλλά και σε δικά μας κρατημέλη ε, μπορεί να χρειάζεται βελτίωση γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν στα κράτη-μέλη και θα πρέπει και πάλι να ξαναρχίσει η κατάρτιση. Η έλλειψη δυνατοτήτων συνεπάγεται ε, ε, κακή χρήση ή ανεπαρκή χρήση των πόρων. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν ε, πάνω από 4% των πληρωμών για το, την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και αυτό το ποσοστό ισχύει για το 2011. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες πόρων. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τέτοιες δυνατότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν γερότερα και ε, καλύτερα ε, τα χρήματα αυτά. Ας δούμε τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τις ειδικέ γι' αυτό ρυθμίσεις. Έχουμε ορίσει 18 προτεραιότητε επενδύσεων που συνδέονται με τέσσερι ε, θεματικού στόχου. Δεν θα τα πω όλα λεπτομερώ, γιατί νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε στι προτάσει. Αν δείτε ε, τους τέσσερις θεματικούς στόχους είναι η πρόθεση της απασχόλησης, η καταπολέμηση της φτώχειας, η επένδυση ε, στην εκπαίδευση και στη διαβίου ε, μάθηση, διοικητικές ε, ικανότητες και δεξιότητες. Αυτή είναι η θεματική στόχη και συνδέονται με θεματικούς στόχους με ευρύτερο ε, ε, πεδίο για την κοινότητα. Δηλαδή η πρόθεση της απασχόλησης σχετίζεται με την ε, βιώσιμη οικονομία, με την οικονομία που έχει σχέση με μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος κλπ. Τα βλέπετε και στα slides αυτά που σας λέω και υπάρχουν και οι τέσσερις θεματικοί στόχοι συνδεδεμένοι με τους βασικούς στόχους πρόθεση της απασχόλησης, κινητικότητα ποιότητα της απασχόλησης συνδέεται με τους στόχους της αύξησης της απασχόλησης το 75% μέχρι το 2020. Ολόκληρη η πρόταση λοιπόν ε, είναι συνεπής εσωτερικά και διασυνδέονται οι διάφοροι στόχοι και θεματικές ενότητες και στο επόμενο slide βλέπετε ότι υπάρχει και η προοπτική του της Ευρώπης 2020. Υπάρχουν συγκεκριμένε διατάξει που διασφαλίζουν ότι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στου άλλου στόχου είναι ανοιχνεύσιμη στο, στη φάση προγραμματισμού και υλοποίηση, ώστε να μπορούμε να λογοδοτήσουμε για το πώ χρησιμοποιούνται τα χρήματα σε κάθε περίπτωση και σε σχέση με κάθε στόχο. Θέλουμε ε, να ε, υπάρχει η υποχρέωση το 60% να σε τέσσερις στόχους προτεραιότητας ε, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, 70% στις μεταβατικές και 80% στις περισσότερο αναπτυγμένες. Δηλαδή όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια περιοχή, τόσο πιο εστιασμένη θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πρόγραμμα. Και εδώ βλέπετε ότι η εκταμίευση ε, γίνεται σε μεγαλύτερο αριθμό στόχων, ενώ πρέπει να εστιαστούμε καλύτερα σε λιγότερους στόχους και αυτή η εστίαση ε, μπορεί να είναι σαφέστερη όσο περισσότερο αναπτυγμένη είναι η χώρα. Μετά από αυτό το slide λοιπόν της συγκέντρωσης σε συγκεκριμένους στόχους, ας περάσουμε σε αυτά που αποτελούν και τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πρέπει η αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών να περάσει σε όλες τις πολιτικές και στον κανονισμό του Κοινωνικού Ταμείου υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση να προγραμματιστούν στοχευμένες δράσεις για την ισότητα ανδρών και γυναικών και τη μη διακριτική μεταχείριση. Δηλαδή υπάρχει και σε γενικό επίπεδο και σε ειδικό επίπεδο και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Άλλο ένα σημείο που κρατάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ότι υποστηρίζουμε την διακρατική συνεργασία. Αυτό έχει να παίξει κάποιο ρόλο και στις εδαφικές προσεγγίσεις, ε, πρωτοβουλίες, ε, τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, ε, θέματα για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρέπει να προωθεί την καινοτομία, δηλαδή χρησιμοποιούμε για την κοινωνική καινοτομία και το πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και μπορούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να το χρησιμοποιούμε για να χρηματοδοτήσουμε δυνατότητες χρηματοδότησης των προγραμμάτων Financial Engineering θα δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λοιπόν, για να δημιουργηθούν πόροι. Μπορώ να δώσω το παράδειγμα των μικροπιστώσεων αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για, την, για να δημιουργηθούν ε, δυνατότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κεφάλαιο κίνησης, ε, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. Με τις προτάσεις μας προσπαθήσαμε όχι μόνο να επεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε σχέση με την τωρινή του μορφή, αλλά να του δώσουμε μια νέα κατεύθυνση ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη συνεργασία με άλλα ταμεία, μεγαλύτερος προσανατολισμός ε, στα αποτελέσματα και απλούστευση όσον αφορά την προσέγγιση του. δεν είναι το πιο εύκολο εργαλείο στη χρήση του. Πρέπει να ε, βελτιωθούν οι γνώσει για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και γι' αυτό θα πρέπει και οι χρήστε του να είναι ενημερωμένοι. Αυτά ως εισαγωγή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μπορούμε να επανέλθουμε στο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. βλέπουμε τη σημασία που έχει η οριζόντια νομοθεσία και η Επιτροπή μας θα πρέπει να τα παρακολουθεί όλα αυτά γιατί πολλές από αυτές τις ιδέες που αναφέρατε υπάρχουν στα βασικά κείμενα αναφοράς. Κατανοώ βέβαια και την σημασία της νομικής βάσης του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κρίμα που ο εισηγητής μας ε, για την οριζόντια νομοθεσία, ο κ. Κωσάνη, δεν είναι παρόν. Όμως η κυρία Μογάν που είναι η εισηγήτριά μας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μπορεί να λάβει το λόγο άμεσα και μετά θα δώσω λόγο στην κυρία Τούρινεν. κυρία Μογά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γενική Διευθυντά, για αυτή την παρουσίαση. Μας δώσατε μία συγκεκριμένη και σαφή εικόνα της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες παρατηρήσεις που έχουν σχέση με τις εργασίες τις οποίες εμείς ήδη ξεκινήσαμε και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στην ομάδα εργασία μας με ε, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα συζητήσαμε αυτό το θέμα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι χαίρομαι διότι η Επιτροπή θέλει να ορίσει ένα ποσοστό του Ταμείου Συνοχής ε, να συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 25% ήδη αποτελεί μια εγγύηση. Ε, κρίμα γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε και μεγαλύτερο. Αρχικά είχαμε μιλήσει για 40% για το Κοινωνικό Ταμείο. και είναι και λίγο σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν χαθεί. Σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο που η απασχόληση είναι κάτι που ανησυχεί και τα 27 κράτη-μέλη, νομίζω ότι εδώ θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο περισσότερο φιλόδοξοι. Ίσως φαίνομαι απαιτητική για το θέμα αυτό, αλλά για την καταπολέμηση της φτώχειας το καλύτερο μέσο είναι η επαγγελματική ένταξη και η κοινωνική ολοκλήρωση. Δεύτερο σημείο είναι το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας που παρέχεται στους απόρους. Έχουμε συζητήσει πολύ το πώς θα μπορούσε αυτό το πρόγραμμα επιστηστικής βοήθειας στους απόρους να διαρθρωθεί και νομικά και πολιτικά. Από όσο θυμάμαι, μιλούσαμε για 84 εκατομμύρια, για, ε, δισεκατομμύρια συγγνώμη, εκ των οποίων τα τρία αφορούσαν, τα 84 αφορούσαν το κοινωνικό ταμείο και τα 3 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούσαν ε, το πρόγραμμα επισητιστικής υποστήριξης των απόρων. Αν μπορείτε να με δώσετε μια διευκρίνηση για το συγκεκριμένο αυτό σημείο, θα σας ήμουν ευγνώμων. Τρίτο σημείο. Σημείωσα αυτό που είπατε για την πολυταμιακή προσέγγιση. Αυτή η πολυταμιακή προσέγγιση έχει μια πολύ θετική πτυχή, στην οποία επιμείνατε, αλλά έχει και μια αρνητική πτυχή. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση της πολλαπλής συμμόρφωσης Ε, είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ναι μεν καταλαβαίνω τους στόχους ε, της ε, δέσμης των έξι μέτρων και ψήφισα υπέρ αυτών, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει και η πολλαπλή συμμόρφωση δεν μας εκπλήσει, αλλά οι πόροι που προορίζονται για την ε, χωροταξία ε, και όπου έχουν αναρμοδιότητα και τα κράτη και οι περιφέρειες είναι ένα θέμα και άλλο θέμα είναι το κοινωνικό ταμείο που πρέπει να ασχοληθεί με κάτι που ωφελεί τους εργαζομένους. Θα το συζητήσουμε στην Επιτροπή μας και θα το συζητήσουμε και με τους εταίρους μας. αλλά το να προσαρτήσουμε το κοινωνικό ταμείο στην πολλαπλή συμμόρφωση μου φαίνεται ότι επιβαρύνει πάρα πολύ αυτούς που ήδη βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσπραγία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προσπαθεί να βοηθήσει αυτούς που βρίσκονται περισσότερο απομονωμένοι και απομακρυσμένοι να βγουν από τη φτώχεια, να βγουν από την απομόνωση. Αν αυτή είναι η προοπτική μας, πώς, να βάλουμε, πώς γίνεται να βάλουμε ένα όριο και να σταματήσουμε αυτή την πολιτική βούληση. Εδώ εγώ βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί μου δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτή η προσέγγιση. Όσον αφορά τις μικροπιστώσεις ε, και τις ε, δυνατότητες χρηματοδότησης, ε, συμφωνώ με την προσέγγισή σας και όντως εδώ υπάρχει πεδίο καινοτομίας. Αλλά νομίζω ότι για τη διαπραγμάτευση αυτής της προσέγγισης δεν πρέπει να υπάρξει κατακαιρματισμός και ως προς τους πόρους και ως προς τα εδάφη. Το είδαμε σε ορισμένες ε, συναντήσεις ε, που είχαμε με την Πρόεδρο. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε τη στρατηγική του, της του 2020 και για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους της Ευρώπης του 2020 μας χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό όραμα και κινητοποίηση και της Ευρώπης και των κρατών με βάση αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, κυρία Τουρίνεν και ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ. Καταρχάς τρία καλά πράγματα και ένα πολύ κακό. Το πρώτο είναι ότι θα θέλαμε να καλωσορίσουμε είναι η απλούστευση. Αυτό το earmarking για το κοινωνικό ταμείο στο συνολικό, στην συνολική προσπάθεια την δημοσιονομική της συνοχή, είναι κάτι το οποίο το εκτιμάμε ιδιαίτερα και χαιρόμαστε επίσης που ευθυγραμμιζόμαστε και με τους στόχους του 2020. Αυτό είναι πολύ θετικό. Σε, για την μακροοικονομική ε, πολλαπλή συμμόρφωση, να επαναλάβω αυτό που είπε και η συνάδελφος, έχουμε μία δέσμη έξι οδηγιών αυτή τη στιγμή, που κατά την άποψή μου είναι πολύ ριζοσπαστική αντιμετώπιση. Ήδη δηλαδή τώρα τιμωρούμε τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τα ελλείμματα και τα χρέη κτλ. Εντάξει, όμως, εάν θέλετε να προσθέσετε και στο κοινωνικό ταμείο ε, και στα ταμεία συνοχής ε, την ε, ε, μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση, τότε τιμωρούμε όχι μόνο τις κυβερνήσεις αλλά και τους πολίτες. Διότι αυτά τα προγράμματα είναι ε, για τα άτομα τα οποία χρειάζονται, ε, χρειάζονται μεγαλύτερη εκπαίδευση, χρειάζονται υποστήριξη, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης σε φτωχές περιοχές της Ένωσης και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα ε, χωρίσετε την Ευρώπη με ακόμα πιο έντονο τρόπο την φτωχή από την πλούσια Ευρώπη. Και η φτωχή Ευρώπη δεν θα μπορέσει ποτέ να ε, ανακάμψει. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο δεν καλωσορίζει τέτοιου είδους μέτρα. Ο κύριος Σερκάσα και μετά η κυρία Χάρκιν και μετά θα σας... θα δούμε ποιος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την, ε, τον Γενικό Διευθυντή για τις εξηγήσεις, για τις εξηγήσεις του. Καταβαίνετε τα Ισπανικά. Επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ Διευθυντά για τις εξηγήσεις σας. Δεν θα σας ε, εκπλήξει το γεγονός ε, ότι θα ακουστούν ε, διάφορα κριτικά σχόλια που απευθύνονται και στον Επίτροπο. Διότι αν θέλετε να ακούσετε τον Ευρωπαίο Επίτροπο, την Ευρωπαίο Πολίτη, συγγνώμη, τις, τους συνδικαλιστές, όλους όσους εργάζονται, οι δικαιούχοι αυτοί που χρειάζονται το ταμείο, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, όλοι όσοι γνωρίζουν ε, πολλές, πολύ δύσκολες ε, συνθήκες διαβίωσης αυτόν τον καιρό, όλοι, όλοι, όλοι αυτοί ασκούν την ίδια κριτική με αυτήν που ακούσατε κι εσείς σήμερα. Όμως μέχρι τώρα δεν ακούσαμε καμία απάντηση από δική σας πλευράς. Ζούμε δύσκολες στιγμές στην Ευρώπη. Και οι πολίτες, πολλοί από αυτούς τουλάχιστον, ζουν κάτω από συνθήκες που είναι, θα τις χαρακτήριζαν δραματικές. Και εμείς εδώ στις Βρυξέλλες θα έπρεπε ενδεχόμενα να ακούμε και τι γίνεται έξω από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι το ταμείο που εξορισμού θα έπρεπε να διορθώσει, αν θέλετε, τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Και ένα μεγάλο μέρος του ταμείου αυτό απευθύνεται στους εργαζομένους. Και αυτούς, τους, αυτούς οι στόχοι θα έπρεπε να μας απασχολούν. Υπάρχουν τα μέσα, αλλά υπάρχουν και οι στόχοι. Υπάρχουν και οι διοικητικέ ανάγκε, δεν λέω, αλλά δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τι διοικητικέ ανάγκε με τι ανάγκε των πολιτών. Και θα έπρεπε εσεί, η κυρία Γενική Διευθυντά ή ο Επίτροπο, δεν ξέρω, θα πρέπει να διευκρινίσετε και στο Συμβούλιο ότι ε, η Επιτροπή μας θέλει να συμμετέχει στην προσπάθεια, γιατί εμείς είμαστε η Επιτροπή που καταλαβαίνει καλύτερα τι συμβαίνει και το Ταμείο δεν μπορεί να ασχολείται με την μακροοικονομία. Ίσα ίσα θα πρέπει να ασχολείται με τις ανάγκες του πολίτη. Μας μιλάνε για τη δημοσιονομική δομή, αλλά δεν μιλάμε για την κοινωνική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Δεν μας ε, μιλήσατε για τις συνέπειες αυτής της περίφημης μακροοικονομικής πολλαπλής συμμόρφωσης, ε, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ε, άνεργοι αυτή τη στιγμή. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα ε, των προγραμμάτων σας στην ε, ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Τα άτομα αυτά δεν δουλεύουν, είναι στην ανεργία, διότι τα κράτη τους δεν μπόρεσαν να σεβαστούν τα κριτήρια τα οποία είχαν τεθεί. Και ε, δεν μπορούν να αναλάβουν ε, ε, οι πολίτες τις ευθύνες των κρατών και το συγκεκριμένο ταμείο, το, ταμείο, ε, το κοινωνικό ταμείο είναι εδώ, δημιουργήθηκε για να καλύψει ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να ή πρέπει να βοηθηθούν. Να ξέρετε πάντως ότι όσον αφορά αυτή τη μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση θα συναντήσετε την αντίσταση του Κοινοβουλίου. Στεναρή αντίσταση, διότι τελικά έχουμε δημιουργήσει ένα τέρας. Δεύτερη ερώτηση, κύριε Γενική, μάλλον τελευταία ερώτηση, κύριε Γενική ε, ε, Διευθυντά. Μία ομάδα βουλευτών και υπαλλήλων που εργάζονται επί τόπου συνειδητοποίησε ποιες είναι, ποια είναι τα αποτελέσματα, συνειδητοποίησαν τα αποτελέσματα της κρίσης. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Όμως, κύριε Γενική Διευθυντά, διαβιβάστε στους ενδιαφερομένους το ότι αντί να πλουστεύουμε να τα πράγματα, θα πρέπει να κάνουμε κάτι για τους γεωργούς διότι επί του παρόντος έχουμε κάποια όργανα τα οποία δεν έχουν καμία ε, εμπειρία, διοικητική εμπειρία και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των γεωργών και κυρίως των ανέργων γεωργών και θα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η χρήση αυτού του ταμείου, τουλάχιστον ε, για αυτούς που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μας ότι τα άτομα τα οποία ασχολούνται με την ε, διαχείριση ε, δαπανούν το 80% του χρόνου τους για να κατανοήσουν τις εντολές των Βρυξελών και οι πόροι δεν είναι και πάρα πολλοί. Αυτοί οι πόροι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να, για να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της κρίσης και να μην ε, ε, δαπανούμε το περισσότερο χρόνο μας ε, για να κατανοήσουμε τα κείμενα για διοικητικές δηλαδή απλώς και μόνο διοικητικές και μόνος διαδικασίες μην καταστρέφουμε τα ίδια μας τα χέρια το έργο μας. Ελπίζω ότι θα ακούσουμε και αυτούς που δουλεύουν εκεί. Γιατί καμιά φορά οι υπάλληλοι εδώ στην, ε, στα θεσμικά όργανα ε, να μην ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, ακούστε και μας σαν Επιτροπή Απασχόλησης που είμαστε κοντά στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει επί τόπου. Και ξέρω ότι υπάρχει μια ασυνεννοησία Ούτε εσείς καταλαβαίνετε τι κάνουμε εμείς, ούτε εμείς καταλαβαίνουμε τι κάνουν οι υπάλληλοι σας. Η κυρία Χάρκιν και μετά ε, θα απαντήσετε εσείς, κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Ένα τεχνικό ερώτημα προς την Επιτροπή καταρχήν. Οι προτινόμενες ε, περιφέρειες μετάβασης. Και αν δούμε τα κείμενα, αν δούμε πώς θα καθοριστούν οι, περιοχές, οι περιφέρειες αυτές, λέει ότι στόχος της νέας κατηγορίας είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση των περιφερειών αυτών, οι οποίες ε, βγαίνουν από τη σύγκληση. Αυτό που ξεχάσατε κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι θα υπάρξουν περιφέρειες, υπάρχουν περιφέρειες των οποίων το ΑΕΠ πέφτει σημαντικά και θα θα κινηθούν προς τα πίσω μέχρι τώρα. Πάντοτε υποθέταμε ότι οι περιφέρειες ε, αναπτύσσονται και ότι οι δαπάνες από τα ευρωπαϊκά ταμεία θα βοηθούσαν σε αυτή την ανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό πράγματι εληθεύει, αλλά τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που ε, το κατακεφαλήν εισόδημα, το ΑΕΠ συνολικά πέφτει και θα υπάρχουν περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία της μετάβασης και επειδή παίρνουμε στοιχεία των του 2007, του 2008 και του 2009 που δεν λαμβάνουν απολύτως υπόψη στα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης γιατί το πλήγμα στο ΑΕΠ έγινε μάλλον το 2010 και το 2011. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία μας ε, ε, θα δούμε δηλαδή τελικά ότι δίνουμε πόρους σε κάποιες περιφέρειες ε, της μετάβασης ε, που δεν το αξίζουν ή που δεν το αξίζουν όσο άλλες και αυτό γιατί βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι οι περιφέρειες πάντοτε αναπτύσσονται. Με κάποιο τρόπο αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη της Κομισιόν. Δηλαδή ποια είναι τα στοιχεία αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η κρίση ή εν περιπτώσει να συσταθεί ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίσει ότι αυτό θα δεν θα παραβλεφθεί. Ιδάλω δεν θα επιτευχθούν σωστά οι στόχοι της πολιτικής συνοχής. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, όπως και η κυρία Μοριντσάρτη θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ υπερψήφισα το Six Pack με κάποιες επιφυλάξεις και ίσως όχι για τους ίδιους ακριβώς λόγους που ε, ψήφισαν οι άλλοι με βαριά καρδιά μερικές φορές πατούσα το πράσινο κουμπί. Πιέστηκα αλλά το έκανα. Παρά τα αυτά θεώρησα ότι ψηφίζουμε κάτι το οποίο σαφώς δεν θα επιλύσει την παρούσα οικονομική κρίση. Ίσως προλάβει κάποια παρόμοια κρίση εύρους και παρομοίου βάθους στο μέλλον. Αλλά από μόνο το αυτό το πακέτο δεν θα λύσει την παρούσα οικονομική κρίση. Το ε, εντάξουμε την πολλαπλή συμμόρφωση του κοινωνικού ταμείου δεν θα βελτιώσει την κατάσταση, για μένα θα την επιδεινώσει. Συμφωνώ λοιπόν με πολλούς από τους προαναλύσαντες σήμερα. Πήγατε πολύ μακριά με την συμμόρφωση όσον αφορά το ταμείο. Και ξέρω ότι το βασικό θέμα είναι η οικονομική διακυβέρνηση, το six-pack, οι κανόνες κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε ε, για ποιο λόγο υπάρχουν και, και τι ελπίζουμε θα πετύχουν αυτά τα ταμεία. Στο νέο πλαίσιο επιδόσεων αναφέρεστε και εδώ θα ήθελα να μου πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Είπατε συγκεκριμένα ότι η Κομισιόν μπορούσε να αναλάβει την διεκπεραίωση των προγραμμάτων και θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες σε περιπτώσεις συγκεκριμένων ε, προβλημάτων ή ελλείψεων κλπ. Αν δείτε κάποιους από τους δείκτες τους κοινή απόδοσης, ανεργία, μακροχρόνια ανεργία και αυτά. Όλα αυτά δεν είναι πάντοτε θέματα που μπορούν να τα ελέγξουν τα κράτη-μέλη λόγω της κρίσης. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τους ανέργους ή τους μακροχρόνια ανέργους, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα των επιδόσεων. Βεβαίως και θέλουμε να χρησιμοποιηθούν τα ταμεία με τρόπο που να βγάλουν 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια και να φροντίσουμε να έχουμε λιγότερα, λιγότερους μακροχρόνια άνεργους. Αλλά στο θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς τη χρησιμοποιούμε. Επίσης υπάρχει μια υπεραπλούστευση. Ε, μιλήσατε για εναρμόνιση των ε, κανόνων. Και τέλος, γιατί αυτό δεν ξέρω τι θα πει, τέλος, γιατί μικροοικονομικά Ζητώ συγγνώμη, λέει ο ομιλήτρια Εντάξει, τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι ακούσατε και τις απόψεις των τεσσάρων πολιτικών ομάδων μέσω των ε, συντονιστών που τις εκπροσωπούν. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο τραπέζης και μετά ε, θα δώσουμε το λόγο σε άλλους, άλλους αντιπροέλους, τον κύριο Τόμας Μάν. Ε, Ευχαριστώ Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πρόταση της Επιτροπής. Μια επίσημη πρόταση που έχει γίνει από την Επιτροπή και η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή. Και υποβάλλεται επί τη βάση λεπτομερέστατων συζητήσεων. δεν ε, έγραψαν την πρόταση αυτή δύο-τρει υπάλληλοι της Επιτροπής. Είναι μια επίσημη πρόταση που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή και τώρα ε, είναι ανοιχτή προς ε, συζήτηση. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά των ερωτήσεων όπως υπευλήθησαν. Καταρχήν, το ποσοστό του 25% με ρωτήσατε αν είναι αρκετά φιλόδοξο είναι φιλόδοξο, διότι και πάλι κινείται ανωδικά. Γιατί είχε μειωθεί. Είχε μειωθεί γιατί αυτό ήταν επιθυμία των 100 μελών. Τα κράτη-μέλη ήταν ελεύθερα να προσδιορίσουν το ποσό χρημάτων που θα ήθελαν να δαπανίσουν για κάθε θέμα και με το πέρασμα των ετών τα κράτη-μέλη επέλεξαν να δαπανούν λιγότερα χρήματα για κοινωνικά θέματα και περισσότερα για δρόμους, τέλο πάντων για επενδύσεις άλλου είδους. Δική του επιλογή ήταν. Δεν ήταν καλή επιλογή, λέει η κυρία Μπεχέ. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει διαφορετική επιλογή, λέει ο μιλητή, και γι' αυτό εμείς βάζουμε αυτό το 25% τώρα είναι ανοιχτό σε πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο βεβαίως και αν δεχθούν τα κράτη-μέλη να φτάσουν πιο πάνω από το 25% εμείς είμαστε ανοιχτοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα ελάχιστο ποσοστό 25% και επίσης προτείνουμε μέσα από αυτό το 25% το 20% τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί για την κοινωνική ένταξη. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο, γιατί στη συνθήκη το κοινωνικό ταμείο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απασχόληση. Και πρέπει να έχει κανείς κατά νου την ερμηνεία και της κοινωνικής ένταξης. Ε, πιστεύει η Επιτροπή ότι μπορούμε να βάλουμε και την απασχολησιμότητα ε, έμεσα στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό γίνεται η πρόταση του να δαπανάτε τουλάχιστον το 20% στην κοινωνική Εντάξει, Θα δούμε αν θα το δεχθούν οι νομοθέτες ως μελλοντική πολιτική. Όσον αφορά την επιστημιστική βοήθεια προς τους απόρους, δεν είναι 3 δισεκατομμύρια, είναι 2,5 δισεκατομμύρια το ποσό που προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Και πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα της πολιτικής συζήτησης που συνεχίζεται. Διαφέρουν οι απόψεις των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι υπέρ του προγράμματος και το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε τμήμα των δραστηριοτήτων τους και άλλα κράτη-μέλη λένε ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση αυξάνοντας ε, ε, το ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης σε μια χώρα για να αποφασίζει ο καθένας αν ε, προτιμά το, το, το ελάχιστο επίδομα που δίδεται σε απόρους να αποφασίζουν ήδη αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για φαγητό ή για κάτι άλλο. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και εξαρτάται αυτό το οποίο θα κάνουμε από την ερμηνεία που θα δοθεί. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί ως επιχειρησιακό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και οι χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και χώρες που δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν μπορούν να δαπανίσουν τα χρήματα σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπήρχε χωριστό κανονισμό για αυτό το θέμα. Πάντω θεωρείται ότι ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πρέπει και πάλι να εξετάσετε προσεκτικά την νομική βάση για να δείτε τι ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά κατά τη γνώμη μας αν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ε, υπάρχει δυνατότητα να γίνει με αυτό το οποίο προτείνουμε. Τώρα για τις παρατηρήσεις ε, σχετικά με τη μακροοικονομική πολυλαπλή συμμόρφωση. Πρέπει να εξετάσουμε στην πράξη πότε μπορεί να εφαρμοστεί, τι συνέπειες θα είχε και τι ακριβώς σημαίνει. Όπως προσπάθησα να εξηγήσω στην πρώτη μου παρέμβαση, δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται στα κράτη-μέλη είναι το τέλος μιας διαδικασίας, δηλαδή έχουν ενημερωθεί τα κράτη-μέλη ότι έχουν ξεφύγει από τους στόχους, ότι πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους κλπ. Και στο τέλος φτάνουμε η συνέπεια δεν είναι ότι παίρνουμε τα χρήματα του κοινωνικού ταμείου και τα δεσμεύουμε. Παραμένουν χρήματα του κοινωνικού ταμείου. Αλλά εάν, παραδείγματο χάρη, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μια χώρα τη σύσταση να δαπανίσει περισσότερα για την ανεργία των νέων και η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη να το κάνει, ενδέχεται να φτάσουμε σε κάποια στιγμή που θα πούμε, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει υψηλή ανεργία των νέων στη χώρα σας και πρέπει τμήμα των κονδυλίων να το χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. σχόλιο της Πρόεδρου εκτός μικροφώνου. Όπως σας είπα, πρέπει ε, να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, γιατί δεν εμπλέκονται οι περιφέρειες σε κάθε περίπτωση. Και αν δώσουμε μια σύσταση σε μια χώρα, θα πρέπει να ε, ερμηνευτεί ω σύσταση προ συγκεκριμένε περιφέρειε όταν συνεργαζόμαστε με περιφέρειες. Επομένω, ε, η πολλαπλή συμμόρφωση δεν σημαίνει ότι μπλοκάρουμε τα χρήματα και τα χρησιμοποιούμε για κάτι άλλο και όχι για για κοινωνικά προγράμματα. Μπορούμε να τα δαπανίσουμε για κοινωνικά προγράμματα. Και θα πρέπει με συγκεκριμένα παραδείγματα να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Για την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει διάφορα πρακτικά σενάρια. Στην παρούσα ε, κατάσταση της Ελλάδας δεν θα ε, εφαρμόσουμε την ε, μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση για την Ελλάδα για τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου. Είπαμε λοιπόν πρέπει να το εξετάσουμε στην πράξη και κατά περίπτωση με συγκεκριμένα παραδείγματα πρέπει να το δείτε. Να μην ε, βάλετε λοιπόν κατευθείαν μια ερμηνεία ε, στη θεωρία. Άκουσα πάντως πολύ προσεκτικά και τα επιχειρήματά σας ε, και τη συγκινησιακή φόρτιση πίσω από τα επιχειρήματα που εκφράσατε. Προσπαθούμε με το Κοινωνικό Ταμείο να κάνουμε αυτό το οποίο κατά περίπτωση είναι σωστό. Δηλαδή τώρα σε περίοδο κρίσης έχουμε προτείνει στα κράτη-μέλη αναπρογραμματισμό αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα πιο γρήγορα ή κάπου αλλού. Τα περισσότερα κράτη-μέλη όμως έχουν βάλει τα χρήματα σε κάποια επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν τόσο ευρύ πλαίσιο που στην πράξη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα ζητάμε συνεργασία για αυτό το οποίο ο πρόεδρος Μπαρόζο αποτελεί πρωτοβουλία για τους νέους. Σαφώς τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κοινωνικό ταμείο και υπάρχει δυνατότητα διότι το 1 τρίτο των χρημάτων που είναι διαθέσιμα για την προγραμματική περίοδο χρησιμοποιούνται και τα υπόλοιπα 2 τρίτα θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει κανείς εστιαζόμενος σε συγκεκριμένους τομείς. Αλλά αυτό απαιτεί δραστηριότητα από τα κράτη-μέλη. Είναι επιμεριζόμενη διαχείριση και η ευθύνη, κατά βάση είναι ευθύνη των κρατών μελών. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε και να κάνουμε ένα προγραμματισμό και με κατεπίγοντα χαρακτήρα εάν χρειάζεται, αλλά να υπάρχει κάποια κίνηση από την άλλη πλευρά, να δούμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ερώτησή σας σχετικά με τις περιφέρειες και για το πώς θα καθορίσει η Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία, πρέπει βεβαίως να είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία αυτά. Σαφώς και θα επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα το Φεβρουάριο-Μάρτιο 2012 σε σχέση με τα δεδομένα του 2010. Επομένως θα υπάρξει προσαρμογή. Παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι το να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτά τα δεδομένα αποτελεί και μια απάντηση σε μια άδικη κατάσταση που υπήρχε στο παρελθόν. Ε, σε περίπτωση που μετακινείται μια χώρα σε διαφορετική κατηγορία. Τώρα εξετάζουμε τις κατηγορίες και προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις αυτές που θα σημειώσει τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Έχω έξω, έξι ομιλητές. Ε, και εδώ πέρα κλείνει και ο κατάλογος και ξεκινάμε τον γύρο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θετικέ εξελίξεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες ε, ανησυχίες. Ε, γι' αυτό θα μιλήσω εν συντομία για την ε, μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση, διότι όπως είπε και είναι απαράδεκτη. Διότι το πρόβλημα είναι να δούμε ποιο χρειάζεται περισσότερο αυτή του είδους την υποστήριξη. Δεν πρόκειται να μπω στις λεπτομέρειες γιατί τα έχουμε ακούσει ακούσει πολλές φορές. Έχω περισσότερες ερωτήσεις όμως. Η υποστήριξη των λιγότερο ευνοημένων ομάδων και η μάχη κατά του αποκλεισμού. Είναι πάρα πολύ καλά πράγματα όλα αυτά πώς ε, βλέπετε να διαμορφώνεται η εφαρμογή. Γιατί είναι πάρα πολύ καλός ο στόχος, αλλά το πρόβλημα είναι η εφαρμογή όλων αυτών. Και χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση και, μια, και την ανάπτυξη ενός διαφορετικού τύπου πρόσβασης και προσέγγισης. Αν θέλουμε πραγματικά να αγγίξουμε αυτούς που χρειάζονται την ε, υποστήριξη αυτή. Ε, εάν εμείς δεν προγραμματίσουμε καλά τις διαδικασίες εφαρμογής τότε πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τα περίπλοκα προγράμματα και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο, στα, ταμεία. Ε, θεωρώ όμως ότι περιοριζόμαστε στις αστικές περιοχές ενώ ε, πιστεύω ότι ε, η, η χρηματοδότηση και η συνδρομή των ταμείων είναι απαραίτητη στην Ήπεθρο διότι εκεί είναι ε, το, το πρόβλημα. Πώς το βλέπετε να διαμορφώνεται όλο αυτό. Επίσης ε, για την πολλαπλή συμμόρφωση σας είπα ότι δεν δεχόμαστε την ε, μακροοικονομική συμμόρφωση όμως άλλες μορφές πολλαπλής συμμόρφωσης χρειάζονται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού. Επίσης αναφέρθηκατε στο mainstreaming στην καταπολέμηση των διακρίσεων Πώς ε, βλέπετε να αναπτύσσεται η πολλαπλή συμμόρφωση στον τομέα αυτό, που δεν θα είναι μακροοικονομική βέβαια. Ο Τόμας Μαν και η μετά η κυρία Γιασούμπλουφσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, η πρώτη σα παρατήρηση ήταν καλή με βάση και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ε, είπατε ότι είναι απλώ πρόταση τη επιτροπή. Είναι πρόταση τη Επιτροπή και αυτή την πρόταση θέλουμε να τη συζητήσουμε. Είπατε ότι ακούσατε τα επιχειρήματα και την ε, συγκινησιακή φόρτιση. Εγώ δεν θα έλεγα συγκινησιακή φόρτιση. Εμείς ε, αγωνιστική φόρτιση έχουμε, γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βλέπουμε ένα ταμείο στο οποίο υπάρχει σαφής ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τα χρήματα αυτά πρέπει να φτάνουν στις ομάδες στόχους, στους δικαιούχους. Δεν είναι λοιπόν συγκινησιακή η φόρτισή μας, αλλά ε, έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις και ξέρουμε ότι αν σωστά χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα θα επιτύχουμε κάτι. Αυτό ήθελα να το πω ως διευκρίνηση. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται κάποιοι πόροι. Ε, ο Αλεσάνδρο βλέπω ότι έχει φύγει από τη θέση, αλλά ήθελα να το πω για να το ακούσει. πρέπει να δούμε τι συμβαίνει επί τόπου κάθε φορά που έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλοι λένε δεν είναι απλές οι διατάξεις. Άλλοι λένε είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πρόσβαση στα χρήματα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να δει κανεί την κατάσταση. Πολύ διαφορετικοί τρόποι να εξηγήσουμε γιατί δεν απορροφώνται τα χρήματα. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να φτάσουμε στις ομάδες στόχους, στους ανέργους, στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Πάντω πρέπει να φτάσουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Και σε ένα σημείο δεν συμφωνώ όσον αφορά το εξαπλό πακέτο και στην ψηφοφορία μπορεί να δει κανείς ποιος ψήφισε υπέρ, ποιος ψήφισε ε, κατά. και δεν συμφωνώ με τον Αλεσάνδρο όταν λέει ότι αυτό το αποφάσισαν οι κυβερνήσει. Τι κυβερνήσει μπορούμε να τι ε, καταψηφίσουμε και στην Ισπανία είδατε ότι έγινε αυτό αλλά μπορούμε και να επιβάλλουμε δεσμεύσεις ε, στις κυβερνήσεις. Έχουμε τρόπους να πούμε ε, στις κυβερνήσεις ότι δεν πρέπει να κατασπαταληθούν τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα τα οποία διατίθενται πρέπει να επενδυθούν με ορθολογικό τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει τρόπος ε, να περάσει αυτό το μήνυμα στους κυβερνώντες. Ξέρω ότι ποτέ δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις όμως και πρέπει να κλείσω με δύο παρατηρήσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία για τους τίτλους των προγραμμάτων όπως έχουμε ε, ε, παραδείγματο χάρη είχαμε το διαβίου μάθηση, μετά είχαμε το Εράσμους. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει το κάθε πράγμα. Όταν λέμε διαβίου μάθηση, αυτό αποτελεί και ένα εμπορικό σήμα θα έλεγα. Δηλαδή η διαβίου μάθηση είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα μήνυμα και τα, τα ονόματα πρέπει να τα κρατήσουμε. Και όταν λέμε Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αυτό ξέρει ο κόσμο και να το κρατήσουμε σαν όνομα. Και άλλο ένα σημείο. Δεν θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένους στόχους, να μην πούμε ευρύτατα γεωργικός τομέας, αλλά να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους ε, για να δείξουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα επιχειρήματα που μας οθούν να υποστηρίξουμε συγκεκριμένο τομέα. Περισσότερη Ευρώπη θέλουμε, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς. Ευχαριστώ κυρία Γιάννη και μετά η κυρία Στάνοβικ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά. Μου αρέσει αυτή η διατύπωση εξυγχρονισμός. του Κοινωνικού Ταμείου μετά το 2013. Όπως όμως και άλλοι συνάδελφοι, έχω και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και έχω και κάποιες απόψεις Θα ήθελα να σας ζητήσω όμως να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια, περίπτωση, σε μια περίοδο κρίσης. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις μας θα πρέπει να είναι άμεσες, κυρίως όσον αφορά την αγορά εργασίας. Μιλήσατε για αυτά τα προγράμματα τα, στα οποία θα δεσμευτούν πολλά ταμεία. Γι' αυτό ρωτώ, θα υπάρχει μια συγκεκριμένη κατανομή, ότι δηλαδή σε κάποιο ε, πρόγραμμα το 25% θα έρθει από το ένα ταμείο, το, το υπόλοιπο από το ταμείο, ας πούμε, ε, το κοινωνικό ταμείο ή το κοινωνικό ανάπτυξης, το ταμείο ανάπτυξης υπαίθρου. Ε, ε, ίσως θα, ίσως, ή μήπως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και μια συγχώνευση των ταμείων. Η κατανομή ε, των πόρων ε, θα μπορούσαν να λάβει, θα μπορούσαν να λάβει υπόψη ε, και κάποιες ομάδες στόχους. Επίσης, μήπως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αλλαγές ενδεχόμενα στις περιοχές που να μείωναν την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης. Άρα θα ανασταλεί η χρηματοδότηση, θα τροποποιηθεί ή τι θα γίνει. Επίσης το αποθεματικό με βάση ποια με ποιες αρχές ε, θα γίνεται αυτό θα καθορίζεται το αποθεματικό με βάση τους υπολογισμούς του κράτους μέλους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί τα όσα προτείνει το κράτος μέλους. Επίσης, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για αυτή την ε, οικονομική, μηχανική ε, μετά το 2013 συνειδητοποιείτε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιείτε πόρους ε, χρηματοδότηση για τους νέους που θα θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το έχετε λάβει αυτό υπόψη σας. Επίσης, όσον αφορά τις αρχές ε, της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να ξέρετε ότι εδώ ε, μας απασχολούν ιδιαίτερα τα κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να αποτελούμε ένα μέρος της λύσης του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση παρόμοια με του προελίσσαντος. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι ε, να καταλάβω αυτό το σημείο όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και σαν μορφή χρηματοδότηση. Μπορείτε να μου δώσετε παραδείγματα για αυτό το financial engineering. Πώ συνδέεται αυτό με του στόχου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εμένα τουλάχιστον δεν μου είναι σαφέ και θα ήθελα περισσότερε διευκρινήσει. Ε, Ντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα εξαρτηθεί από την δυνατότητά του να προσαρμοστεί στα διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται λόγω των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα καλά πράγματα της συμπληρωματικότητας του Κοινωνικού Ταμείου με το ΦΕΝΤΕΡ μέσω της ε, ολοκληρωμένης στρατηγικής με τις ε, στοχευμένους στόχους η καταπολέμηση των διακρίσεων και του, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να στραφεί και για τους άστεγους που πολλαπλασιάζονται σήμερα στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν διαρωτώ με, τι θα κάνετε για τους άστεγους στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του, της, του περιορισμού της εγκατάλειψης του σχολείου, ε, είναι θετικό στόχος γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα ε, κινδυνεύουν να συσσωρεύσουν και τη φτώχεια και την ανεργία. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα όμως τώρα. Ε, υπάρχει έλλειψη όταν ε, συγκεκριμένων λεπτομεριών όταν μιλάτε για το θέμα της φτώχειας. Η, σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απασχολησιμότητα και ε, φτώχεια. Η απασχόληση δεν προστατεύει πια από την φτώχεια. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για φτώχεια, τι, πρέπει να πούμε τι είναι φτώχεια. Σήμερα είναι το 8% στην Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει μια λέξη που είναι πολύ ε, της μόδας χρησιμοποιείται πολύ στην Ευρώπη και αλλού. Κοινωνική καινοτομία. Τι ακριβώς σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνική Καινοτομία. Το λένε πολύ αυτό. Ελπίζω ότι σημαίνει ότι θα δημιουργήσει κανείς ε, μια οικονομία κοινωνική και αλληλέγγυα με όλη την έννοια που έχουν αυτοί οι όροι. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό το, η κοινωνική καινοτομία και θεωρώ ότι το διακύβευμα του να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη είναι προϋπόθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά πρέπει να λάβουμε την κατάσταση που υπάρχει, την πραγματικότητα, τη σημερινή, τα προβλήματα τα οποία δεν εμφανίζονται εδώ. Εγώ λοιπόν θα ήθελα πιο συγκεκριμένα μέτρα και περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Διευθυντά, δεν θα έπρεπε να έχετε αμφιβολία ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Αλλά πρέπει να πω στο πολιτικό προσωπικό που βρίσκεται εδώ ότι πρέπει ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εδώ 13 μέλη. Είναι η πιο σημαντική συζήτηση που κάνουμε. Έχουμε δεσμεύσει και τον Επίτροπο, αλλά δεν είναι λόγος αυτός. Θέλω λοιπόν να πω σε όλους όσοι παρήσανται να κάνουν τη δουλειά τους γιατί αλλιώς δεν, ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ποιο θα είναι η θέση μας στις διαπραγματεύσεις αν δεν είμαστε απολύτως δεσμευμένοι σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει σημαντικότερο θέμα στην ημερήσια διάταξη από αυτό εδώ. Και αν συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε μια γραφειοκρατική ε, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ειδικών, τότε δεν ε, είναι πολιτική αυτή. Αυτό δεν απευθύνεται σε εσά κύριε Γενική Διευθυντά. Ελπίζω ότι το καταλάβατε. Όμως, θα ήθελα να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Φοβάμαι ότι στη συζήτηση αυτή η μακροοικονομική ε, πολλαπλή συμμόρφωση είναι το δέντρο που κρύβει το δάσος. Γιατί βεβαίως είναι σημαντικό αυτό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιείται μια τεχνική την τεχνική Thatcher που θα το έλεγα εγώ, που συνίσταται στο ώστε να επικεντρωθούν όλα σε ένα πράγμα για να μην φανούν τα υπόλοιπα. Αλλά να είστε ε, σίγουροι ότι τα μέλη της Επιτροπής θα τα κοιτάξουν όλα όλα αυτά που θέλετε να δουν, να δουν και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει λοιπόν να σας πω μια σειρά από επιχειρήματα που για μένα κάνουν την πρόταση αυτή απολύτως απαράδεκτη και ελπίζω ότι στο κοινοβούλιο αυτό θα υπάρξει ευρεία κινητοποίηση. Είναι εντυπωσιακό. Θα πρέπει να γίνει μία μελέτη ε, για να δούμε κατά πόσο θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα οποία προτείνεται. Και είναι πάρα πολύ περίεργο το γεγονό ότι δεν έγινε εκ των προτέρων. Η Κομισιόν λέει ότι με αυτό το πακέτο οικονομική διακυβέρνηση, το οποίο δεν ψήφισα, ψήφισα ε, ε, έχουμε προβλέψει κυρώσει για τι χώρε τη Ευρωζώνη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και κάτι αντίστοιχο και για τι υπόλοιπε χώρε. Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω και πάρα πολύ καλά και τι υπόλοιπε Ένωσης. Εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά όλη αυτή τη λογική αν χρησιμοποιείτε τα διευθυντικά ταμεία σαν κρίσιμη μάζα, εισάγετε ε, δυνατότητες ανισορροπίας και ανισότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη που δεν είναι αποδεκτές και που είναι αντίθετες και με, την, ε, με τις συνθήκες. Δηλαδή προβλέπετε μία μάζα με διαφορετική γεωμετρία ε, ανάλογα με τις ανάγκες των κρατών, των κρατών μελών. Δηλαδή ούτως ή άλλως χρησιμοποιούνται δυσανάλογα, μάλλον αντίστροφα από τις ανάγκες τα χρήματα αυτά. Ίσως ε, να, είμαι, να, είμαι, να είναι πολύ καρτεσιανή η λογική μου για να το παρακολουθήσω όλο αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο προβλέπετε, είναι να υπάρχει μια πολιτική σε κεντρικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα ε, η πολιτική αυτή προχωράει προς τις περιφέρειες και είπατε ότι τα πάντα αντιμετωπίζονται μέσα από μια περιφερειακή ε, προσέγγιση. Λοιπόν, τι τιμωρείτε τις περιφέρειες για τις πράξεις ε, ε, των, κρατών μελών. Ε, δεν θα πρέπει τότε να πείτε ότι οι κυρώσεις ε, επιβάλλονται σε επίπεδο περιφέρειας. Τώρα, επίσης λέτε ότι δράτε και ανασταλτικά. Το σύμφωνο σταθερότητας αναθεωρήθηκε, διότι οι κυρώσεις που συμπεριλαμβάνονταν εκεί ήταν αναποτελεσματικές, διότι ήταν απλώς και, και μόνο αποθαρρυντικές, αποτρεπτικές. Λοιπόν, διορθώσαμε το σύμφωνο σταθερότητας και έχουμε κυρώσεις αυτόματες. Τώρα όμως για, το, για τα διορθωτικά ταμεία μας λέτε μην ανησυχείτε, αυτά τα κίνητρα εδώ είναι αποθαρρυντικά. Τελικά τα αποθαρρυντικά τι είναι το αποτρεπτικά κίνητρα, είναι καλό ή κακό. Τη μία φορά είναι καλό και την άλλη δεν είναι. Όντως πρέπει να δείξουμε μεγάλη φαντασία. Αλλά Εφόσον έχουμε να κάνουμε με χώρες ε, που δεν μπορούν ε, να σεβαστούν τα διάφορα κριτήρια λύματος κτλ. Υπάρχουν άλλα μέτρα τα οποία είναι πιο αποτελεσματικά και ίσως κυκλικά αν θέλετε, διότι Πιστεύω τελικά ότι δεν εξετάσαμε αρκετά την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων τύπου υποχρέωση αύξησης των φόρων, ακόμα και του ΦΠΑ, ή στο, και αν δεν είμαι συνήγορος ε, της αύξησης του ΦΠΑ ένα άλλο επιχείρημα στις 21 Ιουνίου όταν η ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, υιοθέτησαν το δεύτερο πακέτο μέτρων για την Ελλάδα θέλαμε να δώσουμε μια ανάσα σε αυτές τις χώρες και επιτρέψαμε να χρησιμοποιηθούν άμεσα τα διαρθρωτικά ταμεία. Δηλαδή έχουμε μια χώρα που έβρισκε στο αδιέξοδο και θελήσαμε να τους, να τους βοηθήσουμε ε, χρησιμοποιώντας με πιο εύκολο τρόπο τα, ε, ε, τα ταμεία. Και τώρα, μερικού μήνε, τρει μήνε μετά, λέμε για τι ίδιε χώρε κόβουμε τα διορθωτικά ταμεία. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Τα διορθωτικά ταμεία είναι ένα εργαλείο πολύτιμο, πάρα πολύ πολύτιμο για, τις, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ προσπαθώ να καταλαβαίνω συνέχεια τι συμβαίνει και τελικά προσπαθώντας να δω τι γίνεται ακούγονται διάφορα ότι χρειάζεται συγχρηματοδότηση, χρηματοδότηση, είναι περίπλοκα, περίπλοκη χρησιμοποίηση του ταμείου. Όμως, όμως, εάν είναι ε, όλοι ειλικρινεί, στο τέλος μαθαίνεις ότι... έτσι όπως ε, θα έπρεπε να λειτουργούν τα διευθυντικά ταμεία, είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει εγώ είναι ότι όταν βομβαρδίζεις ένα παιδί με, με, με, τα με συνέχεια λέγοντας σου τα ίδια πράγματα, κάποια στιγμή γίνεται αυτιστικό και δεν σε ακούει καθόλου. Και ε, από το να χρησιμοποιήσεις το ραβδί και το καρότο, ίσως τελικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε το καρότο και όχι το μπαστούνι. Ε, εδώ έπρεπε ίσω σε διαρθρωτικά ταμεία να σκεφτείτε και κάποια συνοδευτικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη, μια διοικητική υποστήριξη. Ε, ε, με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε. Και όχι να αναγκάζεται το κοινοβούλιο να κινητοποιείται για να βρούμε κάποια στοιχεία στη διαπραγμάτευση. Ζητώ συγγνώμη γιατί μακρηγορώ, αλλά σπάνια μιλάω τόσο πολύ σε αυτή την επιτροπή, τώρα που θέλουμε από τη θέση μου ως πρόεδρος. Τέλος πάντων, να προσθέσω ότι όλοι ξέρουμε πώς ε, αυτή η, και για ποιους λόγους εισήχθη στις διαπραγματεύσεις αυτή η μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση. Τρεις μέρες ε, μετά την ομιλία του Προέδρου Μπαρόζο για την κατάσταση της Ένωσης ε, που προκάλεσε τον θαυμασμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, ενό και ενός τμήματος της Ολομέλειας χωρίς να έχει ενημερώσει τους υπόλοιπους επιτρόπους. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι σωστό σωστό. Ξέρετε, βλέπετε κύριε Γενική Διευθυντά ότι θα έχουμε ε, πολλή συζήτηση ακόμα για αυτό το θέμα. Α, κυρία Πρόεδρε, ε, μερικά δευτερόλεπτα για να συμπληρώσω την ερώτηση που κάνατε και νομίζω θα σας ευχαριστήσω. Το ερώτημα το οποίο ήθελα να θέσω αφορά το, το αποθεματικό επιδόσεων. Και αυτό είναι θέμα παιδαγωγικό. Δεν φοβόσαστε ότι θα οριστούν στόχοι πάρα πολύ χαμηλοί σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποθεματικό, αν θέλετε, ε, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε, παρά να, οριστούν οι στόχοι του 2020. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, για το λόγο για να απαντήσετε, αλλά σύντομα σας παρακαλώ. Ε, Πολύ λίγα έχω να πω για να εκφραστώ ξεκάθαρα μετά από όσα είπατε εσείς, αλλά θα προσπαθήσω. Καταρχήν, δεν ξεκινάμε από το μηδέν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει μια εμπειρία ετών και όπως διαπιστώνουμε, δεν λειτουργήσε πάντοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο για τα κράτη-μέλη όσο και για τις περιφέρειες. Εν γέννη υπάρχει καθυστέρηση στην δημιουργία προγραμμάτων. Τα προγράμματα πολύ συχνά έχουν κάποιο, ένα τεχνητό χαρακτήρα. Και όπως τώρα υπάρχει οικονομική κρίση και όταν λέμε στα κράτη-μέλη, μήπω θα πρέπει να προσαρμόσετε λίγο τι προτεραιότητέ σα, αυτά που θα κάνετε, μα λένε Α, είναι δύσκολο, α προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε απλώ προσαρμογή. Προσπαθούμε να πλαισιώνουμε τα κράτη-μέλη σε αυτή την προσπάθεια. Επισκεπτόμαστε τα κράτη-μέλη, θέτουμε ερωτήσει, προ... Ε, οθούμε προ μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ένα μεγάλο μέρο τη δουλειά του προσωπικού είναι ακριβώς να πηγαίνει σε διάφορες χώρες, να συνομιλεί με τους ανθρώπους και να τους ενθαρρύνει να κινηθούν προς μια κατεύθυνση. Επίσης, όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση, ένα άλλο μέρος μας έχει δεσμεύσει σε ένα ποσοστό σφάλματος ε, που δεν μπορεί να είναι άνω του 2% το οποίο είναι δρακόντιο. Αλλά αυτό οδηγεί σε δράσεις. Εάν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις, ε, στην, κανονική εκ των προτέρων πολλαπλή συμμόρφωση, διακόπτουμε. Και ε, ε, μετά από έξι μήνες, αν δεν υπάρχει διαφάνεια, γίνεται αναστολή για επαόριστον, επαόριστον, μέχρι ότου το κράτος μέλος να έχει δώσει ικανοποιητικές πληροφορίες για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν στο χώρο της πολλαπλής συμμόρφωση. Δεν είναι ότι δεν ε, δεν εμπιστευόμαστε, δεν δίνουμε. Όχι, πηγαίνουμε εκεί, ε, έχουμε συνομιλίες, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τι δεν πάει καλά, γιατί δεν λειτουργεί καλά μια κάποια αρχή, προσφέρουμε τεχνική βοήθεια. Ήδη ε, το θέμα αυτό έχει τεθεί και οι, οι αποφάσεις... Ε, για διακοπή ή για αναστολή ε, επενούνται ιδιαίτερα από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά από την άλλη μεριά μιλάμε για συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό που λέω είναι ότι ποτέ δεν προτάθηκαν ε, οι μακροοικονομική ε, αυτή η πολλαπλή συμμόρφωση για να πληγεί ο τελικός δικαιούχος. Είναι για να εξυπηρετηθεί καλύτερα και να πάνε τα χρήματα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Η πρόεδρος είπε αν δεν υπάρχει, μήπως υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτό και ε, το, ε, σε αυτή τη διάσταση και στη διάσταση της άμεσης επιβολής ποινής. Από τη στιγμή που έχει εισαχθεί στο κείμενο η πολλαπλή συμμόρφωση, δεν λειτουργεί αυτόματα προς το παρόν. Χρειάζεται απόφαση ακόμα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να περάσει κανείς στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες γίνεται συζήτηση και μπορεί κανείς να ε, συνειδητοποιήσει τις πολιτικές συνέπειες. Όμως δεν θα ήθελα να επικρατήσει η η ιδέα ότι ακολουθώ μία μέθοδο θατσερική που δείχνει κάτι για να καλυφθούν όλα τα υπόλοιπα. Όχι. Έχουμε μία μέθοδο η οποία πρέπει να είναι συνεπής και συνεκτική. Ο σκοπός της δεν είναι να τιμωρηθεί ο τελικός δικαιούχος, είναι να βοηθήσει για να υπάρχουν καλύτερα προγράμματα και να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν για να στηθεί στα πόδια της μια χώρα. Για όλες τις χώρες υπάρχουν ε, από θέματα τεράστια για τεχνική βοήθεια. Μερικές φορές υπάρχει υπεροψία, η υπερηφάνεια και οι χώρες δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν όμως ε, χώρες ε, με πρόγραμμα τώρα, αλλά υπάρχουν ακόμα 240 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ε, απομείνει για την οικοδόμηση θεσμικών οργάνων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είμαστε στο 2011. Νομίζω ότι τα προγράμματα είναι σχετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά βεβαίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για αυτό το σκοπό. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε κάποια θέματα που τέθηκαν. Καταρχήν, για την απλούστευση. Ξέχασα τα συγκεκριμένα παραδείγματα απλούστευσης. Πώς η εναρμόνιση μπορεί να είναι απλούστευση. Επειδή υπάρχει διαφορετικός κανονισμός που αναφέρεται στο ίδιο θέμα με διαφορετική ε, με διαφορετική διατύπωση και αυτό μπορεί να δώσει διαφορετικές ερμηνείες σε διαφορετικά μέρη. Δηλαδή βλέπαμε ότι υπάρχει διαφορετικός ορισμός για το ίδιο πράγμα σε άλλο ταμείο από ότι στο κοινωνικό ταμείο. Τώρα προσπαθούμε και να πετύχουμε λιγότερες διαφορετικές ερμηνείες και αποφασίσαμε ότι η προσέγγιση αυτή του ολοκληρωμένου προγραμματισμού θα πρέπει να οδηγεί και σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο λειτουργίας των γραφείων ε, υποστήριξης για να μην λειτουργεί κανείς απομονωμένα αλλά να αντιμετωπίζει μια χώρα ή μια περιφέρεια ολοκληρωμένα. Τώρα το θέμα της, ε, των ονομάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα παραμείνει ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υπάρχουν λόγοι για τον οποίο έχει ε, προταθεί το Erasmus for All γιατί υπάρχουν ε, διάφορα Εράσμους, Erasmus Μούντους, Εράσμους, ε, ε, και μια σειρά από άλλα. Ενώ η διαβίου μάθηση είναι επίσης μια άποψη που ισχύει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως, και εδώ η ιδέα της εναρμόνισης όλων των κανονισμών ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι ενώ ε, μέχρι τώρα λέγαμε «Α, ξέρετε αυτό που ζητάτε είναι ακριβώς εκτός ορίου ε, και δεν μπορεί να ε, καλυφθεί» κλπ. Ρωτήσατε αν δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να ασχοληθεί και με αγροτικά ζητήματα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, το Food for the Deprived, που το πήγαν στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφάσισε. Παρά τα αυτά το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε πολλά κράτη-μέλη για εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα. Αν δεν δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα αυτό μπορεί να μην εξυπηρετούνται πλέον οι άνθρωποι αυτοί. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, γίνεται μια ιδεολογική συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να το φροντίσει αυτό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όσο χωριστό παράθυρο ή ενσωματωμένο στο Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό είναι υποσυζήτηση ακόμα. Αυτή είναι η προϊστορία, αν θέλετε. Επίσης, θα θέλαμε ταχύ αντίδραση από τα ταμεία για την, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Θα μπορούσαν να κινηθούν ε, ταχύτερα από ό,τι διαπιστώνουμε ότι κινούνται τώρα. Και γι' αυτό είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει περίπτωση να δυσκολέψουν την αντίδραση των κρατών μελών ε, οι προτάσεις μας όχι. Αντίθετα, θέλουμε να είμαστε επικεντρωμένοι και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στον τρόπο που αντιδρούν στι εξελίξει στην αγορά εργασία. Δεν βλέπουμε όμω κινήσει προ την κατεύθυνση των προγραμμάτων εκτάκτου ανάγκη. Είναι ένα μηχανισμό που συνεχίζει να λειτουργεί, υπάρχει και τώρα απλώ εφαρμόζεται. Τα αποθεματικά. Τα αποθεματικά είναι αποθεματικά επιδόσεων τα οποία δημιουργούνται σε ένα εθνικό πρόγραμμα. Δεν είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αποθεματικό, υπάρχει σε εθνικό πρόγραμμα. Και, και η χρήση τους προκαλείται από το βαθμό στο οποίο έχει ανταποκριθεί το πρόγραμμα κάποια χώρα. Ε, τώρα, για την ε, ε, χρηματοοικονομική μηχανική και θα επανέλθω και στο δεύτερο σκέλος αυτής της συζήτησης γιατί με ειδοποιούν ότι πρέπει να προχωράω γρήγορα οι άστεγοι. Αυτές είναι κατηγορίες που μπορούν ε, να ενισχυθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δηλαδή το θέμα της απασχολησιμότητας, αλλά τίποτα δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα. Ίσως ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα του, της άμεσης διαχείρισης, το Progress, για να ξεκινήσουμε κάποια πειράματα για να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία. Τα κράτη-μέλη που θέλουν να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά για συγκεκριμένους, σε συγκεκριμένους τομείς έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, να εκπονήσουν τέτοια προγράμματα. Αυτό σε αυτό τους επιστήσαμε την προσοχή. Τους είπαμε ότι μπορούν να ασχοληθούν με θέματα ε, ανεργίας των νέων, για τους αστέγους κλπ. Και τα δύο τρίτα, όπως σας είπα, ακόμα μένουν ε, χωρίς να έχουν δαπανηθεί. Για την κοινωνική καινοτομία θα επανέλθουμε αργότερα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν θέλετε να υπερασπιστώ ακόμα κάποιο σκέλος της ε, δημοσιονομικής πολλαπλής συμμόρφωσης ή αν έχετε ε, φυλάξτε τα κανόνια σας για άλλες φορές <laughs> και θα βρείτε άλλα θύματα. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι, ότι εγώ προτιμώ το καρότο και όχι το μπαστούνι. Γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη και θα πρέπει και εκεί να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να παρουσιάσετε το νέο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και για την κοινωνική καινοτομία και να πατήσετε και στην ερώτηση της κυρίας Ντελή Σα ξαναδίνω το λόγο κύριε Γενική Διευθυντά. Όπως ξέρετε, επί του παρόντος έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Progress. Είναι ένα σχετικά μικρό εργαλείο, αν δείτε το μέγεθος ε, του Κοινωνικού Ταμείου, 76 δισεκατομμύρια, εδώ μιλάμε για 100 εκατομμύρια, όλο μαζί με, την, τα προγράμματα μακροοικονομικής ε, χρηματοδότησης ε, που το υποστηρίζει το ή Κοινοβούλιο και ε, έχουμε το ερώτημα του τι θα κάνουμε στο μέλλον με το πρόγραμμα αυτό. Καταρχάς αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει μια συνέχεια του προγράμματος Progress. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την κοινωνική καινοτομία και μέσω της, ε, του κοινωνικού πειραματισμού. Τώρα το πρόβλημα είναι, το ερώτημα που τίθεται είναι μπορείτε να το εντοπίσετε αυτό, να το αναγνωρίσετε. Εγώ θα δεχόμουν το ερώτημα αυτό από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα πλην των Γάλλων. Διότι στη Γαλλία όντως έχουν κοινωνική καινοτομία που στηρίζεται στην εμπειρία, στα απτά παραδείγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε περισσότερο στην, στις κοινοτικές πολιτικές. Διότι θέλουμε να δοκιμάσουμε νέες εξελίξεις, αλλά θέλουμε να τις, να, τα, να τις δοκιμάσουμε σε διαφορετικές χώρες, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και να διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε ένα νέο όνομα στο πρόγραμμα αυτό και μιλάμε το πρόγραμμα για την κοινωνική καινοτομία και τον εξυγχρονισμό. Αυτό περιγράφει καλύτερα το περιεχόμενο, πιστεύουμε. Ε, ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών, διάλογος, κοινωνικός πειραματισμός, καινοτομία δηλαδή που στηρίζεται στην εμπειρία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο στη χρησιμοποίηση δεδομένων, χρησιμοποιώντας και την, τον κοινωνικό πειραματισμό, διότι πολλές καινοτομίε γίνονται έτσι αυθόρμητα, από ενστικτοδός και δεν υποστηρίζονται από αποδείξεις. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα νέο τρόπο εργασίας. Επίσης θα θέλουμε να συνδέσουμε το πρόγραμμα αυτό με τους βασικούς στόχους του, ε, της Ευρώπης 2020, διότι είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστούν τα πάντα και οι βασικοί στόχοι ε, ακριβώς ε, μας υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουμε. Το να βγάλουμε 20 εκατομμύρια από την φτώχεια, το να συμπεριλάβουμε όλους αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την καινοτομία και τον πειραματισμό. Επομένως, αυτό είναι ο φωτεινός ε, σηματοδότης μας, αν θέλετε, ε, για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. ένα τμήμα, ένα κομμάτι του κεντρικού προγράμματος αυτή τη στιγμή είναι το EURES που είναι ο, ο, σύνδεσμος ανάμεσα στις υπηρεσίες απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή μόνο εξυπηρετεί την διαφάνεια. Δηλαδή να ξέρουμε ποιες είναι οι κενές θέσεις που υπάρχουν σε κάποιες χώρες και να ε, γνωστοποιούμε και μάλλον και να, να, να επιτρέπει την δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων. Άρα αφορά μόνο τη διαφάνεια. Στο μέλλον το Γιούρες θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα και να κάνουμε συνδυασμό. Δεν θα το κάνουμε εμείς βέβαια το συνδυασμό ανάμεσα στις κενές θέσεις ε, και στα βιογραφικά. Δεν θα το κάνουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θέλουμε να το δημιουργήσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι άνεργοι να μπορούν να δούνε κατά πόσον ταιριάζουν με τις απαιτήσει των κενών θέσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις στην Ευρώπη, εδώ και μήνες ορισμένες από αυτές τις θέσεις και δεν μπορούν να καλυφθούν διότι δεν υπάρχει σωστός συντονισμός αν θέλετε και δεν ε, μπορούν να βρεθούν τα απαραίτητα προσό... άτομα με τα απαραίτητα προσόντα. Απ' την άλλη πλευρά είναι περιορισμένη η κινητικότητα ε, του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού ζει σε άλλες ε, χώρες πλην της χώρας του. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο δυνατό τρόπο και πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμα αυτό EURES και να μην περιοριστεί μόνο στη διαφάνεια. Όλα αυτά βέβαια απαιτούν ε, συνεργασία και συντονισμό όλων των υπηρεσιών ε, απασχόλησης στην Ευρώπη. Χρειάζεται τεχνικές ε, προηγμένες όσον αφορά την τεχνολογία γενικότερα ε, θα πρέπει να ε, επενδύσουν αν θέλετε ε, όλες οι χώρες χρειάζεται πολλή δουλειά και στηριζόμαστε τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών απασχόλησης στις, και εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα περνάω στην ε, μακροχρηματοδότηση. Ε, αυτό το macrofinancing ε, μικρό, συγγνώμη, microfinancing δημιουργήθηκε και αρχίζει τώρα τα πρώτα του βήματα. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι προχωρεί πάρα πολύ αργά διότι θα πρέπει να δημιουργηθούν πρώτα τα ειδικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα εφαρμόσουν την μικροχρηματοδότηση. Ε, ξεκινάμε σε αρκετές χώρες και ο αριθμός αυτός των χωρών αυξάνεται. Επίσης είναι σαφές ότι οι διατάξεις αυτές ε, έχουν σαν στόχο την ανέβρεση συγκεκριμένων λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραδείγματο χάρη οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά που δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση αλλού και μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν τις ε, διευκολύνσεις που προσφέρει η μικροχρηματοδότηση. Θα θέλαμε να έχουμε με ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό για αυτή το εργαλείο. Πιστεύουμε όμως ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ε, γι' αυτό χρησιμοποίησα και προηγουμένως το παράδειγμα της οικονομικής μηχανικής. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με την μεθοδολογία που ε, ε, έχουμε επιλέξει για αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η μεθοδολογία και θα να απευθύνουμε έκκληση σε περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμετέχουν, όμως τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να, ε, να βοηθήσει. Αυτές είναι οι εξελίξεις ε, και υπάρχουν τώρα και κάποιες αυτόνομες δημοσιονομικές ε, γραμμές. Είναι λίγο μυστήριες Έχουμε το κονδύλι για τον κοινωνικό διάλογο, για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και τα, τα δημογραφικά και οι οικογένειες των, για τους εργαζομένους. Το τελευταίο, αυτό κονδύλι είναι λίγο, είναι λίγο σαφές. Μιλάμε για σεμινάρια, ε, ε, ε, συνέδρια κτλ. Όμως σε, αυτές, σε αυτά τα κονδύλια προβλέπονται αρκετά χρήματα. Έχουμε τις τομεακές ε, ανταλλαγές απόψεων ε, ανάμεσα στους εργοδότες ε, και τους εργαζόμενους. Και για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, σας έχουμε δώσει και τα ποσά τα οποία συνοδεύουν αυτά τα κονδύλια τα αυτόνομα κονδύλια. Ευχαριστώ. Η κυρία Στάινμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Τον έχουμε ένα πρόγραμμα που θα ασχολείται με την κοινωνική αλλαγή δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακούγεται να είναι καλό, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ε, κατά την ε, κατάρτιση ενός προγράμματος να μην χάνουμε την ποιότητα από το μυαλό μας. Κατά τη γνώμη μου είναι τρία σημαντικά προγράμματα και το καθένα από αυτά έχει πραγματικά τη δική του σημασία. Και γι' αυτό θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση. Σε αυτό το νέο τέταρτο πυλώνα τι, ε, πρόσθετη, τι προστιθέμενη αξία βλέπετε εκτός από την ενημέρωση και την πληροφόρηση γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ποια αλλαγή πραγματικά επέρχεται στα μεμονωμένα προγράμματα και ε, έχω και μια ερώτηση σε σχέση με το ε, EURES που αναφέρατε Υπάρχει και η δυνατότητα παροχής συμβουλών ε, που από τους εργαζόμενους ε, χρησιμοποιείται πολύ. Ε, μερικές φορές δεν είναι αρκετά εκτεταμένη η παροχή συμβουλών. Αυτή η συμβουλευτική θα μειωθεί Και σας υπενθυμίζω και την προηγούμενη ερώτησή μου για την, ε, για τη χρηματοδότησης και την μικροχρηματοδότηση. Αν μπορείτε να μου περιγράψετε με δύο λόγια ε, τι εννοούσατε και στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για τις δυνατότητες Financial Engineering. Ο κύριος Μπουλόν και μετά η κυρία Μόχα. Ε, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερα να πω. Είμαι σκιώδης εισηγητής. Ήθελα να ακούσω την προσέγγιση της Επιτροπής. Προς το παρόν δεν βλέπω την μεγάλη προστιθέμενη αξία για να δανειστώ τον όρο της προηγούμενης ομιλήτριας. Πολλοί από τους, από τους άξονες αυτούς ήδη αποτελούν άξονες τη πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσω πολλών υφισταμένων οδηγιών υπάρχουν. Υπάρχουν τώρα οι γραμμές του προϋπολογισμού για τη βελτίωση της ε, διαφάνειας ε, αυτών των οργανισμών. Δεν διαφωνώ με την πρόταση ενός τέτοιου μέτρου. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις από την Επιτροπή για καινοτομίες μέσω αυτών των εργαλείων. Κάτι τέτοιο θα με ενδιαφέρε περισσότερο. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Να περιμένουμε τις προτάσεις σας και παράλληλα να το σκεφτόμαστε κι εμείς. Η κυρία Μογάν και μετά η κυρία Ντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. μεταξύ των εργαλείων κοινωνικής καινοτομίας ή μεταξύ των προγραμμάτων κοινωνικής καινοτομίας υπάρχει ένα πρόγραμμα για τη συνένωση εργοδοτών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή απάντηση επιτόπου για την απορρόφηση της ανεργίας, κάτι που θα, έδινε, θα αποτελούσε μια πραγματική εξυπηρέτηση για μικρομεσές, για μικρές επιχειρήσεις ε, που βρίσκονται βρίσκονται διάσπαρτες στην περιφέρεια. Ίσως και αυτό αποτελεί και μια απάντηση σαν αυτό που θα περίμενε ο κύριος Μπουλόν που μίλησε προηγουμένως. Θα μπορούσατε να μας πείτε τι πραγματική καινοτομία προσφέρει αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Ντελή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα είναι η θέση των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, διαβάζοντας το έγγραφο, Κάποια σημεία δεν τα καταλαβαίνω. Λέτε κάπου το Progress θα είναι ανοιχτό σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στα μέσα ενημέρωσης. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης, πώς εντάσσονται εδώ. Δεν αναγράφονται οι εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά μιλάτε για τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της αξιολόγησης και ανάλυσης αντικτύπου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται με αυτό το οποίο διαβάζω. Μήπως θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε. Μιλάτε για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε αυτό τον κατάλογο υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι. και αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι η συγχρηματοδότηση φτάνει 15% κατά μέγιστον. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω στη συνέχεια, λέει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Και επίσης να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, πώς θα απλουστεύσετε την αξιολόγηση. Πρόεδρος. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ. Στην κοινή διαχείριση αναφέρεται το EIF. Πώς θα γίνει αυτή η κοινή συνεργασία. Εγώ έχω εξετάσει κάποια προγράμματα μικροχρηματοδότησης ε, και μερικές φορές διαπιστώνουμε επιτυχημένα προγράμματα, αλλά πολλές φορές η βάση είναι πολύ μικρή, δηλαδή η συλλογή εμπειριών είναι πολύ περιορισμένη θα ήθελα να σα ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διαφορά, αν υπάρχει κάποια σύγκρουση ή αν ε, αυτά πάντοτε είναι τα επιθυμητά. Οι περισσότερες ερωτήσεις ε, αφορούν περισσότερο λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσω να ε, ανταπεξέλθω. Θέλω να υπογραμμίσω καταρχήν ότι μιλάμε για μια επέκταση αυτού του οποίου υπάρχει. Δεν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, απλώς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα που να αντικατοπτρίζει αυτό που γίνεται, αλλά να έχει και καινοτομία, αρκετή καινοτομία για το μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Δεύτερον, ποια είναι η αξία του συνδυασμού. Όλοι μας λειτουργούσαμε ε, με βάση οδηγίες κατά την προετοιμασία για απλούστευση και για τη μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση. Και βλέπετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα παράθυρα κάτω από έναν κανονισμό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προσφορά στην γενική αρχή της εναρμόνισης και της απλούστευσης. Ό,τι μπορούσε να ενοποιηθεί το ενοποιήσαμε. Βεβαίως μπορείτε να μας πείτε ότι αυτό είναι κόλπο γιατί τα παράθυρα εξακολουθούν να μένουν χωριστά. Παρά τα αυτά εντάσσονται σε έναν κανονισμό πλέον με μία σειρά ε, στοιχείων. Τώρα, τι έχει γίνει μέχρι τούδε. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κάποιος πειραματισμός. Ας πούμε το EURES. Έχουμε αναπτύξει το δίκτυο το δίκτυο είχε συγκεκριμένο περιορισμένο στόχο. Τώρα εσκεμένα κάτι προσθέτουμε εδώ και προετοιμάζουμε ε, το σύστημα EURES για ε, συγκεκριμένο σκοπό, πράγμα το οποίο στοιχίζει, στοιχίζει και σε ε, εργασία. Οι υπηρεσίες απασχόλησης το έλεγξαν και τους ικανοποιεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουν δουλειά σε ανέργους και δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό σε μια άλλη χώρα και μόνο 2,6% του ε, ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού ζει και εργάζεται σε άλλη χώρα. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις και πρέπει να τις καλύψουμε. Επίσης, να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές, υπάρχει γλωσσικό ζήτημα, υπάρχει η δυσκολία του να μετακινηθεί κανείς σε κάποια άλλη χώρα. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα, ούτως ώστε να συμβεί αυτό. Μια γραμμή είναι θέλουμε να προσθέσουμε μία αντίστοιχη λειτουργία. Αλλά πίσω από αυτή τη φράση, τη, θέλουμε να προσθέσουμε μία αντίστοιχη λειτουργία, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Τώρα, όσον αφορά την γραμμή προπολογισμού για τα πειράματα, ναι, αλλά κάποια στιγμή με τα πειρα... από τα πειράματα πρέπει κανείς να καταλήξει κάποιο συμπέρασμα. Αυτό έγινε και με την περίπτωση της μικροχρηματοδότησης, το microfinance πρέπει κάποια στιγμή να διαπιστώσει κανείς εάν η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ε, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ένα μέρος όμως αυτής της μεθοδολογίας μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερη κλίμακα και να μεταφερθεί ας πούμε στα, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να δημιουργήσει συστήματα μικροχρηματοδότησης ε, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή με το να δημιουργήσει ε, revolving funds για να μην χαθούν τα χρήματα μετά από ένα χρόνο αλλά να ενισχυθούν γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει δυνατότητα κλιμάκωσης ενώ μπορούμε με αυτό, τώρα να κάνουμε νέα πράγματα και να προσαρμοστούμε στις αλλαγές της κοινωνίας. Με αυτό, αυτό θέλουμε να κάνουμε με την κοινωνική καινοτομία. Πολλά είναι τα, ε, τα ζητήματα ε, επί των οποίων θα μπορούσαμε να πειραματιστούμε σε αυτή τη φάση. Δεν θα ήθελα να υπησέλθω τώρα σε λεπτομέρειες. Όλα όσα κάνουμε, όλα όσα κάνουμε στο πλαίσιο αυτού του direct management θα βγει ε, σε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Θα γίνουν πολλές προσκλήσεις ε, στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άρα θα ε, ε, εντοπίζουμε πολύ συγκεκριμένα κάθε φορά τους δικαιούχους. Ε, είπατε ότι υπάρχουν μια σειρά από κατάλληλα πράγματα που μπορούσαν να γίνουν. Δεν μπόρεσα καν να τα καταγράψω όλα όσα είπατε, αλλά πάντως δεν ισχύει ότι ξεχνάμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα ενταχθούν σε αυτές τις προσκλήσεις, θα συμπεριληφθούν σε αυτές τις προσκλήσεις ε, υποβολής προτάσεων. Το ε, η μεγάλη κοινοτομία εδώ είναι ο πειραματισμός. Μην μου πείτε να σας πω συγκεκριμένα σε τι θέλουμε να πειραματιστούμε. Θέλουμε να μας πούν και τα κράτη-μέλη. Πρέπει όμως ε, να, έχουν σχέση με τους βασικούς στόχους της Ευρώπης του 2020 Τώρα για την αξιολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε να γίνει το σωστό είδος αξιολόγησης. Αυτό το οποίο με εντυπωσίασε καθώς επέστρεψα στους τομείς, στο χώρο, είναι η διαφορετική τρόποι χρησιμοποίησης της αξιολόγησης. Κάποιες από τις αξιολογήσεις είναι σε κάποιο έτσι μυστήριο επίπεδο, δεν ε, μας δίνουν στοιχεία και αριθμούς. Εμείς θέλουμε κυρίως στοιχεία και αριθμούς και όχι ε, να ασχοληθούμε θέματα πολιτικής. Υπό την έννοια αυτή πρέπει να, οι αξιολογήσεις να γίνουν επαγγελματικές, να έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πολλές απλώς γράφονται για να υπάρχουν Πρέπει να επανέλθω στο ερώτημά σας για το 15%. Δεν εννοούσαμε αυτό. Αλλά το τι ακριβώς εννοούσατε εσείς, καλύτερα να το συζητήσουμε διμερώς. Δεν έχω να κρύψω τίποτα από τους υπόλοιπους, αλλά θα με βοηθήσει να καταλάβω την ερώτησή σας καλύτερα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Αντίθετα με τις συνήθειές μας, τρία άτομα ζήτησαν το λόγο αφού ολοκληρώσαμε το, γύ, το γύρο των ερωτήσεων. Είναι πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, και μια και έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας και δεν θέλω να δυσαρεστήσω κανέναν, ε, θα τους δώσω το λόγο, αλλά καλό θα είναι να ζητάτε το λόγο εγκαίρως, πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση. Λοιπόν, τρία λεπτά οι ερωτήσεις και δύο λεπτά η απάντηση. Δεν μπορούσα να ζητήσω το λόγο νωρίτερα γιατί ήθελα να σχολιάσω κάτι το οποίο είπατε. Είπατε ότι τίποτα δεν αποδίζει από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα για τους άστεγους. Λέτε ότι τίποτα δεν αποδίζει από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του κοινωνικού ταμείου, τέλος πάντων, ή για, τις, για, την, για μικροχρηματοδότηση κτλ. Όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει δέσμευση από πλευρά των κρατών μελών. Ε, και αυτό το οποίο ρωτώ είναι πώς εσείς προσπαθείτε να, να επηρεάσετε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τους πόρους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να ε, ε, προσανατολίζονται σε αυτούς που τους χρειάζονται, αυτούς που ζουν σε ε, συνθήκες ένδυα. Και δεν πήρα καμία απάντηση σε αυτό το ερώτημα. κυρία Ζίμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που δεν ζήτησα το λόγο νωρίτερα, αλλά νόμιζα ότι θα άκουγα κάποιες απαντήσεις σε προηγούμενες ερωτήσεις. Αλλά όσο περισσότερο ακούω στη συζήτηση, τόσο περισσότερο μπερδεύομαι και δεν έχω καταλάβει ποια είναι η κατεύθυνση, ποιος είναι ο στόχος τον οποίο θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό το πρόγραμμα άκουσα ε, ε, ε, τις ερωτήσεις που παραμένουν και δικές μου ερωτήσεις γιατί δεν έχουν διευκρινιστεί τα θέματα της μικροχρηματοδότησης και των νέων προγραμμάτων κλπ στην ε, Ευρώπη μέσω του EURES θα ε, βρεθούν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, είπατε. Στην Γερμανία έχουμε 2,7 εκατομμύρια ανέργους και εσείς λέτε ότι θα έχουμε 2 εκατομμύρια ε, θέσεις μέσω του EURES σαν στόχο για ολόκληρη την Ευρώπη. Τι είναι αυτό, είναι όφελος και τι θέσει θα είναι αυτές για πανεπιστημιακού, για φουρνάριδες, για μηχανικούς αυτοκινήτων, για βοηθούς, μερικής απασχόλησης, περιορισμένου χρόνου. Δεν θέλω να έχουμε μια μορφή εργαζομένων που θα πρέπει κάθε δύο χρόνια να φεύγουν από, τη θέση, την θέση εργασίας τους και από τον τόπο κατοικίας τους γιατί αυτό δεν είναι η δική μου εικόνα για την κοινωνική Ευρώπη. Ναι. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο και αποτελεί μια καινοτομία διότι από ό,τι φαίνεται δεν ε, συνηθίζεται στην Επιτροπή μας αλλά ε, είναι πολύ ασαφή όλα αυτά τα οποία άκουσα. Μιλάτε για την κοινωνική καινοτομία, για τον κοινωνικό εξυγχρονισμό, μιλάτε για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος. Ε, με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει περισσότερες μελέτες αντικτύπου και συνεπειών και μελέτες εφαρμοστικότητας, αν θέλετε, αυτών των προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης ε, που ζούμε, ε, ε, όταν μιλάμε για καινοτομία και για κοινωνική αλλαγή, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερη κοινωνική σύγκληση σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα έπρεπε να σκεφτούμε περισσότερο. Αυτή η, έλλειψη, η έλλειψη συγγνώμη, εναρμόνισης ή σύγκλησης αποτελεί ένα φρένο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αλλά θα πρέπει και το κοινωνικό ταμείο να ε, χρησιμοποιεί πόρους που να έχουν και μακροοικονομικές συνέπειες. Επομένως, τι είναι αυτό το κοινωνικό ταμείο, κύριε Γενική Διευθύντα, μία, ένα καρότο ή μία καινοτομία. Όχι, μία ανάγκη είναι τι θα τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε την, το επίπεδο δέσμευσης των κρατών μελών. και να σας πω, εμεί ξεκινήσαμε με τους στόχου του 2020, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, να προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Κάνουμε αποστολέ, οργανώνουμε αποστολέ και τους λέμε να υιοθετήσουν ε, προγραμματικά, λειτουργικά προγράμματα. Τους βοηθάμε, τα βοηθάμε τα κράτη-μέλη. Ε, και αυτό δεν γίνεται μία φορά το χρόνο. Αν δείτε τον αριθμό των αποστολών που έχουμε οργανώσει σε κυρίως 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, προσπαθήσουμε να τους ε, αναγκάσουμε να ξοδέψουν κάτι. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν ξοδέψει μέχρι στιγμής το 3% από αυτό που θα μπορούσαν να είχαν δαπανίσει. Βοηθάμε σε τεχνικό επίπεδο, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό ε, ναι, οργανώνουμε αποστολέ. προσπαθούμε να αποτελέσουμε πηγή έμπνευση, να δώσουμε ε, βοήθεια, ε, υποστήριξη καθημερινά στα κράτη-μέλη. Πραγματικά μπορούσα να ε, μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες και να σας εξηγήσω όλα, αλλά από, ε, ε, αλλά από το επίπεδο καθορισμού της πολιτικής μέχρι την καθημερινή, την πραγματικότητα παρεμβαίνουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, σε κεντρικό επίπεδο έχουμε στη διάθεσή μας κάποια χρήματα για να δοκιμάσουμε νέα πράγματα για να προσφέρουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν υιοθετούν δύο-τρία κράτη-μέλη τα οποία συζητάνε παράμερα. Αν θέλουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή κινητικότητα, αυτό θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα προωθηθεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα από τα κράτη-μέλη μόνον. Ε, στο παρελθόν δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Ξεκινήσαμε με το EURES ε, σε εμβριακή μορφή βέβαια, αλλά θα μπορούσε να πείτε ότι δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εμείς πιστεύω ότι το χρειαζόμαστε για να δώσουμε κάποιο νόημα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Θα μπορούσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες και μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το πόσα άτομα είναι εκεί Ξέρω το γερμανικό ενδιαφέρον στο να έχουμε περισσότερους ε, ανθρώπους ε, ε, με τα σωστά προσόντα. Είχαμε και υπουργικές απαφές που μας είπαν ότι υπάρχουν πολλές κενές θέσεις στη Γερμανία που δεν μπορούν να καλυφθούν διότι δεν μπορεί να γίνει ο συνδυασμός με τα κατάλληλα προσόντα. Έστω και αν υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι. Αυτό ακούμε από παντού, ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν τα προσόντα με, την, με, την κοινή, με τις κενές θέσεις. Δεν τα βρίσκω εγώ από μόνος μου, μας τα λένε τα κράτη-μέλη αυτά. Ε, και ελπίζουμε ότι το 2012 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και θα, μετά θα ε, έχει τη δυνατότητα όλη η Ευρώπη να έχει ένα σύστημα ταξινόμησης ε, ε, των προσόντων και των αναγκών και των προσόντων και των γνώσεων που απαιτούνται. Ε, ο βασικός στόχος του εργαλείου αυτού είναι να υπάρχουν χρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαθέσιμα έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το, αυτός ο πειραματισμός, αυτή η καινοτομία που θα, που θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Και αυτό είναι ο μόνος λόγος ύπαρξης. Τώρα βέβαια βασικό να σας πω, ε, βασικό να σας πω, ε, που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει ορισμός ε, σταθερός για την κοινωνική καινοτομία, διότι η πειραματισμό διότι αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λέει η Πρόεδρος.